Okay, ladies and gentlemen, colleagues, can I bring... Αγαπητοί και κύριοι, ας ξαναρχίσουμε για το απόγευμα. Έχουμε τρεις εκθέσεις να εξετάσουμε σήμερα. Λευκή βίβλος για το μέλλον των μεταφορών πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τον εισηγητή κύριο Γκρός. Ευχαριστώ πρόεδρε λευκή, λευκή ρίβλος, που έχουμε λάβει και από που αποτελεί βάση για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Και που θα συζητήσουμε με αρκετά χρόνο στη θέση μα, όχι υπερβολικό, επί τη βάση των προτάσεων τη Επιτροπή πιστεύω ότι μπορεί να μας επιτρέψει και μάλλον οφείλουμε χάρη σε αυτή να προχωρήσουμε το χύτερο δυνατό σε συγκεκριμένες προτάσεις και να τη χειριστούμε με όσο δυνατόν πιο ρεαλιστικό και πραγματιστικό τρόπο. Λευκή βιβλός ή λευκή βιβλός αυτή δεν είναι η πρώτη. Γι' αυτό θα ήταν καλό ίσω να στρέψουμε το βλέμμα προς τα πίσω και να κοιτάξουμε τι έχει γίνει και στο παρελθόν ως προς ε, τους στόχους που είχαν οριστεί, κατά πόσον επιτεύχθηκαν ο περιορισμός του, των εκπομπών του οξυδίου του άνθρακα, ο εξυγχρονισμός τεχνολογικός, η ιστορική του εξωτερικού κόστους, όλα αυτά λοιπόν γιατί δεν επιτέχθησαν. Είναι γιατί οι στόχοι δεν ήταν αρκετά σπουδαίοι ή γιατί δεν είμαστε σε θέση να του επιτύχουμε. Και δεύτερον, η λευκή αυτή βίβλος εξετάζει δίνει προτάσεις για την περίοδο μέχρι το 2030 περίπου. Δεν είναι κακό πράγμα βέβαια, αλλά ω έχει τώρα η κατάσταση και από την εμπειρία που έχουμε συλλέξει του τελευταίου μήνε σχέση με το Συμβούλιο, η περίοδος αυτή, ο ορίζοντας αυτός ο μπορεί να είναι και επικίνδυνος. Διότι για το κατά πόσο θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς και πώς. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι να διατυπώσουμε συγκεκριμένου ρεαλιστικού στόχου από πλευρά του Κοινοβουλίου, να επικεντρωθούμε περισσότερο σε μια περίοδο 10-15 ετών, χωρί να λησμονούμε και την παραπέρα περίοδο, με συγκεκριμένε προτάσει για τι οποίε μπορεί το Κοινοβούλιο να αξιοποιήσει για να εκφράσει τι προσδοκίε του είχαμε πράξει, είχαμε δώσει βασικές ιδέες, όπως την αποτελεσματική συλλειτουργικότητα ως, προϋπολο, προϋπόθεση για συνδυασμό με στόχο πάντα και με γνώμονα τον άνθρωπο αλλά και την οικονομία τον συνδυασμό κάθε μορφής μεταφορών με βάση τις δυνατότητες και τεχνολογία και την κατάσταση των μεταφορών που υπάρχουν ή την, περι, την περιοχή και με πτυχές βέβαια οικονομίας, περιβάλλοντος αλλά και ασφάλειας και εναρμόνισης. Αυτός ο στόχος καθίσταται νομίζω πολύ σαφές μέσα στο έγγραφο που έχουμε να εξετάσουμε. Θα μπορούσε όμως να υποστηριχθεί και να υπογραμμιστεί ακόμη περισσότερο για την πρώτη περίοδο 2010 τα επόμενα 10-15 χρόνια. Και έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να ορίσουμε όχι μόνο στόχους και ποσοστά, αλλά και συγκεκριμένε χρονολογίες ο στόχους. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αυτό που είχαμε ορίσει στόχο 2005 δεν επιτευχθεί εγκαίρως. Άρα μπορούμε να ορίσουμε πιο συγκεκριμένους στόχους για τον περιορισμό και τον εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, με συγκεκριμένες ε, πρωτοβουλίες, πρακτικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να ήταν ε, για μένα μια πρώτη προσέγγιση. Το άνοιγμα των αγορών για το οποίο είμαστε καταρχήν ε, σύμφωνοι, αλλά σύμφωνοι για μια ορθώς λειτουργούσα αγορά, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί η αγορά να απελευθερωθεί πάση θυσία και με οποιαδήποτε προϋπόθεση. Ήταν αυτό που είχαμε δει και σε σχέση με το καμποτάζ πριν από μερικά χρόνια. Το κοινοβούλιο δηλαδή θέλει να προχωρήσει στην απελευθέρωση αγοράς χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μπορούμε να δεχθούμε την παρέτηση από ορισμένους συγκεκριμένους όρους και κανόνες που θα πρέπει να ισχύουν για να λειτουργεί σωστά αυτή η αγορά. Αυτό πρέπει να το καταστήσουμε ακόμη πιο σαφέ, πιστεύω, σχέση με τόσο προτείνει το έγγραφο. Συγκεκριμένη και ρεαλιστική στόχη για μένα είναι επίση να μπορούμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα σε σχέση με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Είδαμε από το μέχρι τώρα διάλογο και τώρα το θέμα που μας απασχολεί στον τομέα, ιδιαίτερα το συνδρομικό, ότι πάντοτε εμείς Μιλούμε στο Κοινοβούλιο ξεκάθαρα και με ευρύς πλειοψηφίες διατυπώνουμε στόχους, τόσο οικονομικούς όσο και στόχους με χαρακτήρα που χαρακτηρίζουν και προσανατολίζουν την, Επιτροπή, την πολιτική των μεταφορών, αλλά αυτούς τους στόχους όχι μόνο τους παραγνωρίζουν, αλλά επιπλέον ε, λαμβάνονται και αποφάσεις οι οποίες Ε, έχουν επιπτώσεις κοινωνικές σε σχέση με τις θέσεις εργασίας τις οποίες τα κράτη-μέλη προβάλλουν ως επιβαλλόμενες ε, αρνητικές επιπτώσεις της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν, εφόσον δεν το πράττουν οι άλλοι, το Κοινοβούλιο να καταστήσει απόλυτα σαφέ ότι θέλουμε μια ανοιχτή αγορά, μια αγορά η οποία πρέπει να λειτουργεί με συγκεκριμένου κανόνε, αλλά μια ανοιχτή αγορά που δεν μπορεί να έχει χώρο ούτε για εργασιακό ντάμπινγκ, ούτε για περιβαλλοντικό ντάμπινγκ, ούτε για υποβάθμιση των αξιών που για μα είναι σημαντικέ. Εάν δεν έχουν αντίρρηση, συνάδελφοι, μπορούμε στα θέματα αυτά της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, στον χώρο των μεταφορών, να ε, ετοιμάσουμε ένα έγγραφο μεθοδικό, ένα έγγραφο ε, συνοπτικό επίσης, το οποίο όμως θα προτείνει συγκεκριμένες ε, προτάσεις και πρωτοβουλίες που περιμένουν από την Επιτροπή για το μέλλον. Ένα ε, έγγραφο, το οποίο φυσικά μπορεί να στηριχθεί σε, αυτό, σε αυτή τη λευκή βιβλίο που είναι πολύ καλή βάση, όπως είπα, για την προοπτική του 2050 εν γέννη, αλλά ιδίω για τα προσεχή 10-15 χρόνια. Χαίρομαι λοιπόν πολύ για την συνεργασία με τους συναδέλφους εδώ στην Επιτροπή. Ελπίζω ότι μπορούμε να προσβλέπουμε σε μια περαιτέρω καλή συνεργασία και θα έχουμε ένα πολύ καλό κείμενο για την πολιτική των μεταφορών στο «Είναι Ευρώπη στο μέλλον». Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρός. Η κυρία Γέγκερα από την Κομισιόν πρωτού δώσω το λόγο στους Ευρωβουλευτές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαι. Κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, Καταρχήν θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να ευχαριστήσω την Επιτροπή Τραν για την ε, συνεχή υποστήριξη της προς την Κομισιόν κατά την προετοιμασία της ε, Λευκής Βίβλου. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ματιό Γκρός ε, για όλη τη δουλειά που έχει κάνει εκείνος, ξεκινώντας από την έκθεσή του και την, ανακοίνωση, την έκθεσή του για την ανακοίνωση για έναν βιώσιμο χώρο μεταφορών το 2009. Η Λευκή Βίβλος υιοθετήθηκε στις 28 ε, Μαρτίου. Ο ε, Αντιπρόεδρος Κάλλας ε, σας την παρουσίασε και έκτοτε είχαμε πολλές ευκαιρίες να τη συζητήσουμε. Η Λευκή Βίβλος προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον και γενικά οι αντιδράσεις που έχουμε λάβει μέχρι τώρα είναι γενικές. Είναι θετικέ. να δράξω την ευκαιρία να σα ενημερώσω ότι πριν λίγε μόλι ημέρε οι Υπουργοί Μεταφορών στο Συμβούλιο συζήτησαν το ίδιο θέμα και να σας ε, παραθέσω τι λένε. Ε, επικροτούν το, τη Λευκή Βίβλο, σημαντικό κείμενο το οποίο ε, συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα του τομέα, στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, στους περιβαλλοντικούς στόχους. Τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι κατάλληλη βάση για την ανάπτυξη μελλοντικών μέτρων στον τομέα της πολιτικής μεταφορών. Ε, μπορεί οι πολιτικοί και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι να έχουν ε, ε, διστάμενε απόψεις σε κάποια θέματα, αλλά χαιρόμαστε που βλέπουμε μια αυξανόμενη συνένεση όσον αφορά τον εντοπισμό των προκλήσεων και την ανάγκη για μέτρα και για τις γενικές γραμμές δράσης που διαγράφονται. Αυτό έχει να κάνει ότι οι στόχοι της πολιτική ε, μεταφορών, ε, περιβάλλοντος ε, και κοινωνικοί στόχοι συνδέονται μεταξύ τους. Είναι απαραίτητο να μειωθεί το κόστος των καυσίμων, όπως επίσης είναι απαραίτητο να καταπολεμηθεί η αλλαγή του κλίματος και να μειωθεί η παγκόσμια ρήπανση. Οι τεχνολογίες που μπορούν να κάνουν βιώσιμες τις μεταφορές είναι και αυτές που θα βοηθήσουν τις βιομηχανίες μας να είναι ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά. Ε, αυτό θα είναι ωφέλιμο και για την κοινωνία και θα μειώσει και το κόστος ε, της ε, συμφόρησης για τις διάφορες επιχειρήσεις. Σημαντικό είναι να υπάρχουν συνδυασμένε μεταφορές και να υπάρχουν ποσοτικοί στόχοι σχετικά με τις δράσεις. Η Ρευκή Βίβλος προσπαθεί να πετύχει τον συνδυασμό των διαφόρων τρόπων μεταφοράς και θα θυμάστε ότι το 2001 ζητήσαμε για ζητήσαμε αυτό το συνδυασμό των διαφόρων τρόπων μεταφορών. Το 2011 θέλουμε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή ε, αυτής. Ε, χρειάζεται λοιπόν περισσότερη αποτελεσματικότητα. Κάθε τρόπο μεταφορών θα πρέπει δηλαδή να μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο φορτίο, να γίνεται μεγαλύτερη χρήση των ε, σιδηροδρόμων καθώς και των πλοίων. Ωστόσο, ε, θα συνεχίσουν και οι οδικέ μεταφορέ. Είναι λοιπόν σημαντικό να ασχοληθούμε με τη διαφοδιαστική και τι καλύτερε τεχνολογίε. το σύστημα μεταφορών θα πρέπει να ε, ε, βασίζεται σε ένα, ε, ενωμένο, ε, ένα ολοκληρωμένο δίκτυο, όχι σε συνδεδεμένα μεταξύ τους εθνικά δίκτυα. Ο κύριος Γκρός αναφέρθηκε σε αυτά στην έκθεσή του και θα πρέπει να επικεντρωθούμε ε, στην ε, βελτίωση του συστήματος μεταφορών. Θέλουμε λοιπόν χρήση όλων των ε, τρόπων μεταφοράς ώστε να έχουμε βιωσιμότητα και να μπορέσουν οι πολίτες μας και οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν το δικαίωμα στις μεταφορές. Στόχος είναι να επιβεβαιώσουμε αυτό το δικαίωμα και να δημιουργήσουμε μια πολιτική η οποία να ε, λαμβάνει υπόψη τις ε, κοινωνικές, ε, οικονομικές και, περιβαλλοντικές, ε, και τους περιβαλλοντικούς στόχους. Επίσης θα εξεταστούν οι δυνατότητες μείωσης των μεταφορών χωρίς όμως να προβληθεί ευμερία. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας να πω ότι έχουμε 40 δράσεις τις οποίες ε, θα προτείνει η Επιτροπή για τα επόμενα 10 χρόνια και ελπίζουμε εντός της παρούσας θητείας. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι δράσεις αυτές και ευθυγραμμίζονται με την φιλοδοξία των στόχων αυτών. Για παράδειγμα, για τους σιδηροδρόμους προτείνουμε ε, να ανοίξουν οι εσωτερικές ε, αγορές για, για τις μεταφορέ, μεταφορές, ε, ολοκλήρωση των υποδομών. Όσον αφορά την τεχνολογία, θέλουμε μακροπρόθεσμους φιλόδοξους στόχους για πρότυπα ενέργειας για όλα τα οχήματα και θέλουμε επίσης περισσότερες ε, προϋποθέσεις ε, για την ε, χρήση, για την απορρόφηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να αποφύγουμε στρεβλώσεις λόγω φορολογίας και να εξεταστεί και το θέμα της φορολογίας των οχημάτων των επιχειρήσεων. Εάν αυτές οι πέντε δράσεις Εάν πέντε από τις 40 δράσεις που προτείνουμε εφαρμοστούν, τότε θα πλησιάσουμε πάρα πολύ ε, τις ε, σημαντικές αλλαγέ που θέλουμε να πετύχουμε στον τομέα των μεταφορών. Κάποιοι θα μιλούσαν για επανάσταση. Ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηρίξει τη στρατηγική μας και τις προσπάθειές μας και ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε τους κοινού μας στόχους. Ε, ε, όσον αφορά την μετατροπή των στόχων σε πρόγραμμα εργασίας θα συζητηθούν κατά τη συνάντηση του Σεπτεμβρίου. Προσβλέπουμε στην ανταλλαγή ε, απόψεων μαζί σας ε, για την Λευκή Βίβλο που πιστεύουμε ότι αποτελεί κοινή προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. much, Ευχαριστώ πολύ κυρία Γέικερ. Θα δώσω το λόγο στις πολιτικές ομάδες. Ε, πρώτα η κυρία Σεναλόβα για, τη για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι το 2050 αποτελεί σημαντικό έγγραφο το οποίο ε, καθορίζει τις ε, μελλοντικέ κατευθύνσεις ε, στην πολιτική μεταφορών αλλά και σε άλλους τομείς ε, πολιτικής. Ε, το, δεν ασχολείται μόνο με τον τομέα της ενέργειας, ε, έχει να κάνει και με το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την ασφάλεια. Η ασφάλεια για μένα είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες. θα θυμάστε και την έκθεση που υιοθετήσαμε σήμερα το πρωί. Γι' αυτό βλέπω τη Λευκή Βίβλο όχι μόνο ως βάση για την συζήτησή μας, αλλά και ως σημείο εκκίνησης για ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε ρεαλιστικά και αποτελεσματικά μέτρα μέχρι το 2020. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι βήματα προβλέπει η Κομισιόν. Η Λευκή Βίβλος βασίζεται σε προηγούμενα έγγραφα, τη Λευκή Βίβλο του 2001 και την ε, αξιολόγηση που έγινε το 2006. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίζεται στο, στην έκθεση για το μέλλον των μεταφορών του 2010. Όλα αυτά τα έγγραφα ε, θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στη Λευκή Βίβλο συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης σχετικά με το κατά πόσο ε, έχουν ε, επιτευχθεί οι στόχοι του 2001. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τους παλιούς στόχους οι οποίοι ισχύουν ακόμα, θα πρέπει όμως να προσθεθούν και νέοι. Η Λευκή Βίβλος αποτελεί μοναδική ευκαιρία να δημιουργηθεί ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος μεταφορών, ο οποίος ε, θα συμπεριλαμβάνει 27 κράτη-μέλη, τα οποία όμως έχουν διαφορετικά σημεία κίνησης. Αυτό αποτελεί σημαντική πρόκληση διότι το επίπεδο των υποδομών και των υπηρεσιών μεταφορών ποικίλει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ξέρω ότι η Λευκή Βίβλος ε, τονίζει το θέμα αυτό και το εκτιμώ. Θα πρέπει να έχουμε εργαλεία ευρωπαϊκής πολιτικής ε, που να ε, ενθαρρύνουν την σύγκληση στα κράτη-μέλη. Στο, στο τομέα αυτό θα πρέπει το έγγραφο να είναι πιο συγκεκριμένο. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ο συνδυασμός των διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Αυτό θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις και ε, σημαντική χρηματοδότηση. Η Λευκή Βίβλος θα πρέπει να αποτελέσει τρόπο ε, συνδυασμού των διαφόρων ε, μεθόδων μεταφοράς και όχι να συμβάλλει στην ανταγωνιστικό, στον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Επίσης, η Λευκή Βίβλος είναι πολύ φιλόδοξη και Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη δυνατότητά τους ε, να πετύχουν τους στόχους. Καθότι όμως ε, δεν είναι βιώσιμη η παρούσα κατάσταση, ε, συμφωνώ με την θέση της Λευκής Βίβλου. Η Λευκή Βίβλος προτείνει 10 βασικούς στόχους. Υπάρχει όμως ένα αλλά. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση σχετικά με την επικουρικότητα όσον αφορά τις αστικές μεταφορές καθώς και την ε, χρήση ε, ε, αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα στα κέντρα των πόλεων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποιο πλαίσιο θα πρέπει να υπάρξουν κάποια εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ίδιο ισχύει και για άλλους στόχους, όπως είναι η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Άλλη σημαντική πτυχή είναι η εσωτερική αυτή του εξωτερικού κόστους και η αρχή του ότι ο ρηπαίνων πληρώνει. Οι ίδιες προϋποθέσεις θα πρέπει να ισχύουν όσον αφορά τα τέλη και τους φόρους που θα επιβάλλονται σε διάφορους ε, τρόπους μεταφοράς. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε εκφράσεις όπως είναι η χρήση των τεχνολογιών και η αποφυγή ε, περί των μετακινήσεων. Η Λευκή Βίβλος επίσης αναφέρεται στις ε, ευκαιρίες εργασίας και στις ε, συνθήκες εργασίας. Ο τομέας αυτός ε, απασχολεί 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όσον αφορά την ποιότητα των ε, θέσεων εργασίας, ε, την επαγγελματική κατάρτιση. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να καθορίσετε καλύτερα η κοινωνική πτυχή. Είμαι σίγουρη ότι η βιωσιμότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών ακολουθούν το ένα το άλλο. Είμαι λοιπόν ε, υπέρ οποιοδήποτε μέτρο που θα βελτίωνε ε, την ε, τις υπηρεσίες για τον χρήστη. Η συμπεριφορά του χρήστη, του, του επιβάτη, είναι πολύ σημαντική. Συμφωνώ λοιπόν με οποιαδήποτε πληροφορική εκστρατεία για το θέμα αυτό και επίσης ένα απλό συμπέρασμα. Οι δημόσιες μεταφορές είναι ε, σημαντικό στοιχείο για τη μακροπρόθεσμη πολιτική μεταφορών στην Ευρώπη και είναι απαραίτητο ε, να εφαρμοστεί αυτή σε ευρωπαϊκό, ε, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάισνερ για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι βέβαια οι μεταφορές ε, με πολλές, από πολλέ απόψει πολύ σημαντικέ για την Ευρώπη, αποτελούν βέβαια τη πολυδελική στήλη ε, της τη οικονομία μα, ταυτόχρονα είναι ε, και μεγάλη πηγή εκπομπών και γι' αυτό είναι στόχο περιβαλλοντικό για μα. Και πιστεύω θα πρέπει ένα έγγραφο που κοιτάει στο μέλλον των μεταφορών να προσπαθήσει να συγκεράσει αποτελεσματικές μεταφορές, καλές μεταφορές και σε αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Γκρός που θα επιτρέπουν την πρόσβαση στους πάντες σε όλα τα μέσα αλλά και από ταυτόχρονα θα υπηρετούν όλους τους στόχους που έχουμε ορίσει ως προς το περιβάλλον, την ασφάλεια, την πρόσβαση για τους πιο ηλικιωμένους, δικαιώματα των επιβατών και ούτω καθεξής. Είναι πολλοί οι στόχοι που έχουμε προσδιορίσει. Και φυσικά αυτό προποθέτει και μια διαρκή προσαρμογή, μετάλλαξη με βάση και τις ισχύουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες. Δεν μπορούμε δηλαδή τώρα καν να διανοηθούμε τι θα υπάρχει το 2050, αν θα υπάρχει NFS σύστημα μεταφορών, αν υπάρχει σύστημα παροχής υπηρεσιών στον επιβάτη που, ή στον οδηγό που ε, θα μας προσφέρει δυνατότητες που δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί αυτή τη στιγμή. Επίσης θα πρέπει να αναζητηθεί η πιο αποτελεσματική λύση. Εδώ πρέπει να ομολογήσω ότι δεν συμφωνώ πάντοτε με τις προτάσεις της Επιτροπής. Αντιλαμβάνομαι ότι κάνει προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ποσοστά, τι ποσοστό μέχρι πότε, μέχρι το 2030 Φερρυπίν 30% από τις οδικές μεταφορές στα... Ε, στους σιδηροδρόμους ή τις ε, πλωτές μεταφορές πάνω από 300 χιλιόμετρα και το αντίστοιχο, σε αντίστοιχε συνθήκες αργότερα για 50% ποσοστό. Αλλά αυτό δεν μπορεί να ισχύει συλλήφθη. Δεν μπορούμε να λέμε ότι σε κάθε περιοχή, κάθε περιφέρεια οι μεταφορές που θα ξεπερνούν τα 300 χιλιόμετρα θα πρέπει κατά 30% να έχουν μεταφορτωθεί μέχρι το 2030 στο ε, χώρο των σιδηροδρομικών μεταφορών των πλωτών. Πρέπει να δούμε τι συνθήκε επικρατούν και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτή η μετακύληση και γι' αυτό καλό θα ήταν οι ποσοστιαίες αυτέ μονάδε να αντιμετωπίσουν ω γενικέ προτάσει. Επίση, έγινε μια επίσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα της ε, ομάδα μα, τη επιτροπή μα. Ε, όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε και τις, τις πλωτές μεταφορές εσωτερικών υδάτων, που ε, βέβαια ήξερα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η μέθοδος και οικολογική μέθοδος οι πλωτές μεταφορές και δεν θα πρέπει να τις εξετάζουμε σαν ευκαιρία οικολογική και οικονομική μόνο για αποστάσεις άνω των 300 χιλιόμετρων μπορούμε και για μικρότερες αποστάσεις κατά τρόπο αποτελεσματικό, οικονομικό και οικολογικό να, και καθαρό να ε, αξιοποιήσουμε τις πλωτές οδούς ε, σε κάθε περίπτωση. Επίσης, ένα ενιαίο πολύ λειτουργικό δίκτυο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασφαλώς είναι μια καλή ιδέα, αλλά δεν πρέπει και να λησμονώσουμε ότι μπορεί να έχουμε τριλειτουργικούς διαδρόμους έτσι ώστε να μπορεί κανείς κατά τρόπον απρόσκοπτα, αποτελεσματικό συμφέροντα οικονομικά και οικολογικά να μεταπηδά από το ένα, από το ένα, μέσο μεταφορών στο άλλο. Και ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι μπορούν να εξελιχθούν περισσότερο οι ιδιωτικέ ιδιωτικές μεταφορές περαιτέρω, χάρη στην εξέλιξη τεχνολογίας και προς ε, λύσεις πιο οικολογικές ε, Επίση, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα τρόπο τιμολόγηση και έκδοση των εισιτηρίων για τι μαζικέ μεταφορέ, ο οποίο θα εξυπηρετεί τον πελάτη, τον επιβάτη, θα διευκολύνει εκείνον που έχει δυσκολίε, θα του καθοδηγεί προ πιο αποτελεσματική χρήση των μεταφορών. Φερρυπίν, εάν το διαδίκτυο δεν μπορεί να μου δώσει πληροφορίε, όπω λέω πάντα, πώ θα ταξιδέψω από τι Βρυξέλλες για τη Μαδρίτη, συνδυάζοντα το τρένο, το αυτοκίνητο, το λεωφορείο και ούτω καθεξής, ε, θα καταλάβω ότι μόνη μου και η πιο απλή λύση να πάρω το αυτοκίνητο και να πάω κατευθείαν. Ε, αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επίσης θα πρέπει να δούμε με, με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ε, ομολογών για ευρωπαϊκά σχέδια για επενδύσεις ε, ή με βάση την στήριξη που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε τέτοια εγχειρήματα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για την πιο ορθολογική ανάπτυξη των μεταφορών, αλλά πάντοτε μονόδος ότι πρέπει αυτές να παραμείνουν αποτελεσματικές και ουσιαστικές. Ευχαριστώ κύριε Ζάτπορ για ε, εκ μέρου της ομάδας του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και επιστρέφουμε στη βάση, θα έλεγα. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών, έναν ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών. Και αυτό για να βοηθήσουμε στην εξυπηρέτηση της νέας αγοράς. Αυτή για μένα είναι η προστιθέμενη αξία μιας ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών. Και τίποτα παραπάνω. Ως προς αυτό λοιπόν, το λευκό βιβλίο που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι κατά κάποιο τρόπο είναι καλό, αλλά εν μέρη. Σίγουρα συμφωνώ με κάποια από αυτά που ήδη υπόθηκαν για το γεγονός, ας πούμε, ότι δεν μπορείς ε, με ρεαλιστικό τρόπο να μειώσει την κινητικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό που έχουμε στο Λευκό Βιβλίο σε κάποιο βαθμό, Πρόεδρε, είναι ένα μείγμα ε, πρακτικών ζητημάτων με θεωρίες. Μιλά για μεγάλα οράματα, για κάποια πράγματα, ενώ για άλλα πράγματα μιλά για πολύ πρακτικές πτυχές της πολιτικής αυτής. Ως προς αυτό, λοιπόν, αυτό που πιστεύω ισχύει είναι ότι πολλά από αυτά τα, τις θεωρίες και τα οράματα ε, είναι στην ουσία ε, θεωρίες όπως σας είπα πριν από 40 χρόνια το 1970, τη δεκαετία του 70, όπως και οι περισσότεροι από εσά θα θυμάστε, αυτό το είδος τα οράματα, τα έγγραφα για τις μεταφορές που βγαίνανε στη δεκαετία του 70, ότι θα πετούσαν τα αυτοκίνητα, από το Λονδίνο στο Σίδνεϊ θα φτάναμε σε 45 λεπτά και κοιτάξτε πού έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. <coughs> Και αυτό είμαι λίγο διστακτικό σε σχέση με αυτέ τι ε, προβλέψει για τα επόμενα 40 χρόνια. Είναι τελείως εκτός πραγματικότητας Τώρα, ήθελα να μιλήσω πιο συγκεκριμένα για κάποιες από τις προτάσεις. Καταρχήν, αυτή η πρόταση για τα αυτοκίνητα έξω από τις πόλεις μέχρι το τέλος αυτής της περίοδου. Μα είναι ανοησία τέτοια. Ε, εντάξει, μιλάμε πάλι για την τιμολόγηση των δρόμων και δήθεν θα αλλάξουμε τις συνθήκες, με τις, μάλλον τις συνήθειες του κόσμου. Αυτά είναι κοινωνική ε, κοινωνικό μαγείρεμα. Στην ουσία χρειάζεται να αφήσουμε την αγορά να διαχειριστεί τα πράγματα. Μιλάμε σε μια άλλη φάση για την σταδιακή εξάλληψη των συμβατικών αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούν μάλλον συμβατικά καύσιμα. Εντάξει, μπορεί να έχουμε σε κάποια στιγμή στο μέλλον ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί με την σύνδεξη, με την ενέργεια από τη σύνδεξη, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο για την ώρα, οπότε θα αφήσουμε κατά μέρος. Από την άλλη πλευρά, συμφωνώ με τις προτάσεις της Κομισιόν και την ουσία αυτών των προτάσεων για το πώς θα κατευθύνουμε ένα μικρό κονδύλι στη βελτίωση των, μετα... των μεταφορών. Δηλαδή, να κοιτάξουμε πού υπάρχει συμφόρηση, πού υπάρχουν ώρες αιχμή μέσα στο πλαίσιο του συστήματος, και φυσικά συμφωνώ και για τα θέματα του ενιαίου εναέριου χώρου. Αξίζει τον κόπο να το προωθήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και συμφωνώ και για το συντονισμό της χρηματοδότησης, γιατί το είπαμε και παλαιότερα, ότι ε, περνάμε μία περίοδο μεγάλων περιορισμών και από ό,τι προβλέπετε θα συνεχίσει να ισχύει αυτό για το εγγύς μέλλον. Ας βασιστούμε λοιπόν σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μα και ας μην σκεφτόμαστε ότι μπορεί να έχουμε ένα πίθμενο πηγάδι από το οποίο θα βγάζουμε διαρκώ χρήματα. Τέλος, Πρόεδρε. Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία για αυτό το λευκό βιβλίο. Υπάρχουν και πολλά σημεία στα οποία διαφωνά και διαφωνώ κατ' ουσίαν. Ε, πρόκειται για την αγορά, για ολοκλήρωση και βοήθεια προς την ε, ενιαία αγορά, αυτά και τίποτα παραπάνω. Κύριε Κράμερ. Όταν ο κύριος Πράτπρον ε, λέει ότι ε, η αγορά ε, καθορίζει όλα αυτά, τότε συμφωνώ, αλλά έχει καταστραφεί αυτό στις μεταφορές λόγω της πολιτικής βούλησης. Δεν δίνουμε χρήματα στους σιδηροδρόμους ώστε να είναι πιο ακριβή. Έχουμε υποχρεωτικά ειδικά διόδια για, τα, για τους συνδρόμους, ενώ οι οδικές μεταφορές είναι πολύ πιο φθηνές. Είναι τελείως τρεβολωμένη η αγορά και ακριβώς γι' αυτό έχουμε το αποτέλεσμα. Έχουμε κάποιους γενικούς στόχους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές. Εγώ υποστηρίζω ότι χωρίς ε, αλλαγές στους τρόπους μεταφορών ε, δεν θα, δεν θα πετύχουμε το στίχο αυτό. Οι μεταφορές ευθύνονται για το 30% των εκπομπών πολύ χειρότερο είναι ότι από το 1999 έχουν αυξηθεί ε, οι εκπομπές κατά 35% στον τομέα των μεταφορών, ενώ στους άλλους τομείς έχουν πέσει κατά 10%. Το οποίο σημαίνει ότι ε, αυτό που έχουμε πετύχει με ε, δισεκατομμύρια ευρώ των φορολογουμένων από μείωση το έχουμε αντισταθμίσει με αύξηση στον τομέα των μεταφορών. Η Γερμανοί κάνουν πολιτική χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ε, τις μεταφορές. Από το πρωτόκολλο του Κιώτο είχαν αποκλειστεί οι μεταφορές παρότι είναι μια από τις χειρότερες πηγές ε, εκπομπών και γι' αυτό είναι θετικό το ότι έχει αναγνωρίσει η Κομισιόν ότι χωρίς ε, τροποποιήσεις, χωρίς αλλαγές στον τρόπο μεταφορών δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Υπόθηκε ότι από 300 χιλιόμετρα και πάνω ε, θα πρέπει να, να υπάρξει αλλαγή στις μεταφορές, αλλά υπάρχουν ε, και, και μικρότερες αποστάσεις για τις οποίες δεν χρειάζεται να γίνει καμία τροποποίηση. Ο ε, Επίτροπος Κίνοκ ήθελε να, μεταφορεί, να, μεταφέρει τις μεταφορές από το δρόμο στους δρόμους. Αυτό δεν το απέτυχε και στην αξιολόγηση του, της Λευκής Βίβλου ε, δεν αναλύθηκε γιατί δεν έχουμε πετύχει το στόχο αυτό. Ε, απλά εισάγαμε τον όρο του commodality των συνδυασμένων μεταφορών ε, Γι' αυτό επικροτούμε ότι σε τούτη την Λευκή Βίβλο ότι έστω και με καθυστέρηση, έστω και με παράκαμψη, επασχετώσει θέλουμε την μεταφορά των μετακινήσεων στους σιδηροδρόμους και στις θάλασσες. Αρνητικό είναι ότι η τελευταία δήλωση της, Επιτρο... της Κομισιόν ότι τα 10 χρόνια ε, θα πρέπει να γίνουν ε, ε, θα πρέπει να επιτευθούν οι στόχοι, αλλά από το 2013 και μετά θα έχει λήξει η θητεία των επιτρόπων, οπότε δεν θα του ενδιαφέρει η πλήρωση των στόχων πια. από το 2030 μέχρι το 2005 ε, πρέπει να έχουμε μείωση 5% δηλαδή 5% το χρόνο. Αλλά εγώ ξέρω πολύ καλά ότι όποιος δεν ξεκινήσει σήμερα δεν θα πετύχει ούτε τον στόχο του 1% τον χρόνο, πόσο μάλλον ε, ε, το 20% μέχρι το 2020. Πρέπει να ξεκινήσουμε ήδη σήμερα για να πετύχουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους. Εάν ε, επί 20 χρόνια δεν κάνουμε τίποτα και μετά περιμένουμε ότι η λύση θα έρθει από τον ουρανό, μόνο οι εκπομπές θα έρθουν από τον ουρανό, κατά τα άλλα τίποτα. Αυτό θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντική αδυναμία. Επίσης, εάν ε, πετύχω το, στό, τους στόχους μου μέχρι το 2030 και πάλι δεν ε, θα αναφέρουμε, δεν θα αναφερόμαστε στο στόχο του 1990, θα είμαστε ακόμα 8% πάνω από, τον, από το επίπεδο του 1990. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος αυτός ε, δεν είναι καθόλου φιλόδοξος. Επίσης έχουν παραλυφθεί κάποια πράγματα, για παράδειγμα η αποφύγη μετακινήσεων. Οι πράσινοι λένε αποφυγή των ε, μεταφορών, ε, αναδιάρθρωση. Ε, ενώ λέτε ότι με, κανέναν τρόπο δεν θα αποφύγουμε τις μεταφορές. Αλλά βλέπουμε... Βλέπουμε για παράδειγμα μεταφορά ψαριών από την, Φιλανδία, από την Σκανδιναβία στην Ασία και μετά πίσω στη Σκανδιναβία. Ε, αλλά όλα αυτά είναι εις βάρος των φορολογούμενων ε, και του περιβάλλοντος. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να αποφύγουμε τις περιττές μεταφορές και θα πρέπει να εξετάσουμε και τις συνθήκες πλαίσιο. Ήδη αναφέρθηκε σε αυτές. Εάν δεν αλλάξουμε τις... Ε, ε πλαίσιο δεν θα πετύχουμε τίποτα και το, το έχω ξαναπεί οι μεταφορές στην Ευρώπη παρά είναι φτηνές Για παράδειγμα, έχουμε δημιουργήσει αυτοκινητόδρομους στην Ισπανία με δισεκατομμύρια των φορολογούμενων, αλλά... Ε, διόδια υπάρχουν στον αυτοκινητόδρομο ενώ δεν υπάρχουν στους τοπικούς ε, δρόμους και έτσι όλος ο κόσμος χρησιμοποιεί τους ε, τοπικούς ε, δρόμους και υπάρχει εκεί μεγάλη συμφόρηση. Εάν λοιπόν δεν αλλάξουν οι συνθήκες πλαίσιο δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας. Κλείνοντας, να πω ότι είναι καλή η πρόταση αυτή αλλά θα πρέπει να την βελτιώσουμε πάρα πολύ. Εάν δεν αλλάξουμε την διατύπωση δεν θα αλλάξουμε ούτε τις μεταφορές. Θέλουμε να βελτιώσουμε ε, το περιβάλλον για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Κάνσια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ε, εισήγηση σε αυτό το μεγάλο θέμα που νομίζω θα πρέπει να μας συμφιλιώσει με ένα μεγάλο όνειρο στην ουσία διατηρώντας αυτά που υπάρχουν, ε, τις υπάρχουσες υποδομές δηλαδή και την κρίση που μας ε, στραγγαλίζει εδώ και κάποιο καιρό. Αυτή είναι η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή να έχουμε αυτό το μεγάλο όραμα για το 2050 και μεγάλους σπουδαίους στόχους, αλλά ταυτόχρονα προσπαθήσουμε αυτά να τα προσαρμόσουμε στη σημερινή πραγματικότητα ενώπιον της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε, διότι δεν δουλεύουμε με βάση το λευκό βιβλίο, αλλά με βάση το πραγματικό οικονομικό πλαίσιο. Αυτό θα πρέπει να είναι η προσπάθεια που θα καταβάλουμε εμείς. Και τα λέω αυτά γιατί το να κοιτάμε μπροστά είναι σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να φτάσουμε και ζωντανοί εκεί, γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε τη ζωή μας στον δρόμο. Γιατί πιστεύω πως η κατάσταση οικονομική ε, στην οποία βρισκόμαστε θα την ε, περιέγραφα ως λίγαν δραματική. Και θα πρέπει να δώσουμε και κάποια μηνύματα, κάποια σημαντικά μηνύματα ήδη από τώρα. Να συνοψίσω σε πέντε σημεία τα όσα θεωρώ μπορούν να είναι αυτοί οι στόχοι, κύριοι στόχοι. Πρέπει να μιλήσουμε για μια ανάπτυξη των βιώσιμων μεταφορών και ήδη με αυτά τα λόγια έχουμε θέσει τις τρεις προϋποθέσεις ώστε να καταστούν βιώσιμα, δηλαδή οικονομική βιωσιμότητα που είναι ε, όχι όπως παλαιότερα στην πρώτη θέση, βιωσιμότητα κοινωνική και περιβαλλοντική. Πρέπει να απομακρυνθούμε από το πετρέλαιο, να κάνουμε σημαντικές αλλαγές και η υπερνική ενέργεια περνά κρίση, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ε, Ένα σώρο εναλλακτικέ λύσεις θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα Δεύτερη πτυχή είναι η πτυχή της απελευθέρωσης, γιατί αν δεν μιλάμε για ανοιχτό, ανοιχτή αγορά, αν και ρυθμισμένη, ο Γκρός το τόνισε καλά, όχι με κάθε κόστος βέβαια, αλλά με κάθε κόστος θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ελεύθερη αγορά με τους ίδιους κανόνες για όλους. Και έπειτα θα το συζητήσουμε και στο επόμενο θέμα που αφορά τους σιδηρόδρομους. Ενιαίος δηλαδή Ευρωπαϊκός Χώρος Μεταφορών που περιλαμβάνει τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ουρανό, το ε, ενιαίο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά αυτό ο ενιαίο χώρος να συνδέεται και με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό θα πρέπει πάντα να το έχουμε υπόψη μας. Αυτό σημαίνει ανταγωνιστικότητα στην αγορά. Τρίτη παρατήρηση είναι η... ο συνδυασμός των διαφόρων τύπων μεταφοράς, γιατί αν δεν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ε, και να ενεργήσουμε σωστά για τις ροές και τους κόμβους με σωστό τρόπο, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Και έπειτα έχουμε και το θέμα του πότε και με ποια χρήματα, γιατί είναι δύο σημαντικέ πτυχέ, οι οποίε όμω δεν μα απασχολούν πάρα πολύ μέχρι στιγμή. Καλά έκανε ο Γκρό και κοίταξε για το πιο κοντινό όριο των 10 ετών, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε ει βάθο ε, την κατάσταση PPP, ορθολογισμό των θεμάτων. Αυτό θα πρέπει να είναι το πιο σημαντικό σημείο για να δοθεί μια απάντηση σε αυτή τη δύσκολη φάση που διανύουμε. Ευχαριστώ. Ο, Ο κύριος Αλκαντράου. Τέσσερα λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ξεκινώ με τον εισηγητή. Τον ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του θέματος. Είμαι ε, βέβαιος ότι θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία στο μέλλον. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι δεν μπορώ να ακολουθήσω στη σκέψη του κύριο Μπράντμπερν. Μπορεί να έχουμε την τάση να προάγουμε την ελεύθερη αγορά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποτελεί την πανάκια και ότι με το που θα απελευθερωθεί ο τομέας των μεταφορών θα επιτυχθούν αυτομάτως όλα τα προβλήματα. δεν θα έχουμε τα υψηλά ποσοστά της ναι. μεταφοράς στις ε, οικολογικές και οικονομικές μεταφορές είτε των φορτίων είτε των επιβατών μέχρι το 2040 εάν δεν προσέξουμε και δεν σχεδιάσουμε προσεκτικά το σύστημα αυτό. Χαιρό λοιπόν για τις προτάσεις. Θα ήθελα ωστόσο να διατυπώσω και κάποιες επικριτικές παρατηρήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων που προτείνονται αφορούν το δεύτερο τμήμα της περίοδου. Εγώ θα ήθελα η δική μας Επιτροπή να ασχοληθεί με τις προτάσεις και την υλοποίηση των μέτρων στο πρώτο χρονικό, στην πρώτη χρονική περίοδο, μέχρι το 2015-20 το πολύ. Και φυσικά τα πάντα θα εξαρτηθούν από την πολιτική βούληση των κρατών μελών. Εάν αποδειχθεί ότι υπάρχει η βούληση να γίνει υποχρεωτική η εσωτερική των εξωτερικών ε, δαπανών, ε, εφόσον το θελήσουν δηλαδή οι κυβερνήσεις, πολύ καλά, αλλά έχω πολλές επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό. και το Συμβούλιο, το ΣΥΠΗΝ, την προηγούμενη εβδομάδα ε, έκρινε εντό εισαγωγικών θετικά όλα αυτά τα μέτρα, όλε αυτέ τι προτάσει. Αλλά δεν θέλω να δω πολύ συγκεκριμένα όταν έρθουν στην ουσία του τα μέτρα και η εφαρμογή του πώ θα αντιδράσει το Συμβούλιο. Επίση, στα οικονομικά. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε το πώς η κινητικότητα και η αναδιαμόρφωσή της θα χρηματοδοτηθούν. Θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός για την μετάβαση στο σιδηρόδρομο, επί παραδείγματι, ένας μηχανισμός που θα εξασφαλίζει την χρηματοδότηση αυτής της μετάβασης και ούτω καθεξής. Και επίσης, ήθελα εν συντομία να πω ότι διάφορες παράγραφοι ή κεφάλαια των προτάσεων θα πρέπει να ε, συμπεριλαμβάνουν πάντοτε και τις κοινωνικές, τα κοινωνικά μέτρα. Ο εργαζόμενος Φερρυπίν. δεν λαμβάνεται υπόψη επαρκώς στον χώρο των ε, μεταφορών. Και εκεί ασφαλώς θα πρέπει να ενσωματωθούν μέτρα τα οποία θα ε, ισοδυναμούν με, θα έχουν στην συνέπεια την προστασία των κοινωνικών συνθήκων. Επίσης, στις, ε, στον περιορισμό των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα μπορεί να είναι φιλόδοξες οι προθέσεις, αλλά μιλισμονούμε ότι τις αρμοδιότητες στον τομέα αυτό δεν τις έχει στα χέρια της η Επιτροπή, αλλά τα κράτη-μέλη. Σε ποιο βαθμό λοιπόν μπορούμε να τα επηρεάσουμε. Δεν Έχουμε να επιλύσουμε ένα ε, γόρδιο δεσμό. Και επίσης, θέματα όπως η καινοτομία στο χώρο της μεταφοράς επιβατών, ηλεκτρικά λεωφορεία και άλλα ζητήματα. Πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λεπτομερέστερα εν την πορεία. Ευχαριστώ. Κυρία Σάρσαρ, πρόεδρε ευχαριστώ, θα είμαι όσο δυνατόν πιο σύντομη. Αντίθετα με άλλους ομιλητές θεωρώ ότι το όρομα και η φιλοδοξία που παρουσιάστηκε είναι ευπρόσδεκτα. Δεν μπορούμε να τυπώσουμε επικρίσει γιατί δεν υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα δράσεω και δεν έχουν ληφθεί οι δεσμεύσει ούτε καν στον δημοσιονομικό τομέα. Η εκπρόσωπο τη Επιτροπή μα είπε ότι υποστηρίζουν ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο των μεταφορών μάλλον παρά το συνδυασμό διαφορετικών χώρων των μεταφορών των κρατών μελών επιμέρους. Πολύ καλή ιδέα αυτή λοιπόν. Και πολύ καλή ιδέα. Να μην λησμονηθούν οι περιοχές που απέχουν κάπως από το κέντρο της Ευρώπης. Είπα επίσης ότι πρέπει να έχουμε πολύ συγκεκριμένα προγράμματα δράσης και ιδέες για τη χρηματοδότηση, διότι ξέρουμε πολύ συχνά το Συμβούλιο δεν την ειδικών ους σε αυτά τα σχέδια, όσο φιλόδοξα και ωραία και να είναι. Και μπορεί και να μην υλοποιηθούν ποτέ. Ευχαριστώ κύριε Φόσνερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα σίγουρα να συμφωνήσω με κάποιες από τις παρατηρήσεις του συναδέρφου κυρίου Μπράτμπορν. Σίγουρα είναι αλήθεια να πούμε ότι υπάρχουν εδώ κάποιες λογικές λύσεις και καλές πρακτικές τις οποίες θα πρέπει να εξετάσουμε. Ωστόσο, το έγγραφο αυτό φαίνεται αφελές σε κάποια σημεία του, παρουσιάζει τη γενική ιδέα, εάν εξετάσει κανείς πιο προσεκτικά το κείμενο, Όταν διαβάζω πιο προσεκτικά το κείμενο, αρχίζω και αναρωτιέμαι. Αν κοιτάξουμε το κοινωνικό θεματολόγιο στους διάφορους τρόπους μεταφοράς. Για παράδειγμα, για τους εργαζόμενους εκεί, την κοινωνική ατζέντα για τις ναυτιλιακές μεταφορές, ε, για τις υπεύθυνε αερομεταφορές. Ε, τι συζητάμε εδώ πέρα. Έχουμε και τη Γενική Πρωτοβουλία 2011. Ε, Εγώ δεν επιδιώκω τις κακές συνθήκες εργασίας σε καμία εταιρεία και σε κανέναν τομέα. Ήμουνα συνδικαλιστρία στον ε, τομέα αερομεταφορών επί πολλά χρόνια. Ωστόσο, όταν διαβάζω αυτό εδώ πέρα, φαίνεται σαν η σαν να μην υπάρχουν ε, καθόλου ε, σχετικές διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συλλογικέ συμβάσει ε, και φαίνεται σαν η Ευρωπαϊκή Ένωση να πρέπει να ε, ασχοληθεί με τέτοια πράγματα. Πάντως, ε, επιφανειακά διαβάζοντα το, δεν ε, φαίνεται πολύ καλό. Επίσης, όσον αφορά τις ε, πρωτοβουλίες για την ασφάλεια, νομίζω θα πρέπει να εξετάσουμε τις καλύτερες πρακτικές. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τα νομικά δεσμευτικά μέτρα. Στο σημείο 16, το για την οδική ασφάλεια και το Zero Vision. Ε, δεν ξέρω ποιος θα αποφασίζει ε, ποιο, ποιος τραυματισμός είναι, ε, ποιος είναι ελαφρά τραυματισμένος και ποιος όχι. Ε, γενικά τα διαβάζω αυτό και αναρωτιέμαι ποιος θα αποφασίζει τι είναι τι, πόσο πολύπλοκα θα πρέπει να είναι, πόσο πολύπλοκες θα πρέπει να είναι οι διατάξεις όσον αφορά την ε, μεταφορά επικίνδυνων ε, υλικών, ε, την πρωτοβουλία 20. Έχουμε κάποιες διατάξεις σε εθνικό επίπεδο, θα εμείνουμε σε αυτές ή θα έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες. Γενικά θα πρέπει να εξετάσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών, το σημείο 21, νομίζω ότι έχουμε αρκετά δικαιώματα επιβατών για να μας κρατήσουν για όλη μας τη ζωή. μετά από την ηφαιστειακή στάχτη, μήπως πρέπει να ε, ε, ξανακοιτάξουμε την κατάσταση στον τομέα των αερομεταφορών. Θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη μας το κόστος για τους διάφορους τομείς. Και τέλος, ναι, έχω στηρίξει το ΣΕΖΑΡ. Θα πρέπει οι κυβερνήσεις να το υποστηρίξουν αυτό ό,τι αφορά την, ε, ε, τη διαμόρφωση των τιμών κλπ. Αλλά όταν μιλάμε για νέο ε, δίκτυο χρηματοδότησης θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κοιτάξει τι προϋπολογισμό έχει και πώς δαπανεί τα χρήματα, διότι δεν υπάρχουν πρόσθετα χρήματα. Και κύριε Πρόεδρε, τέλος, όσον αφορά την ευφυγή διαμόρφωση τιμών και τη φορολόγηση. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα. Είναι πολύ ε, γενικό το κείμενο και δεν θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε τις αγορές ε, των ασφαλίσεων. Νομίζω θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Ε, κάπως ανησυχητικά μου φαίνονται όλα αυτά, αλλά ναι, υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία. Σίγουρα υπάρχει περιθώριο για διευκρινήσει. Ε, φαντάζομαι και για διαφορετικές απόψεις. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντυρό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να εκφράσω την ευχαριστησή μου για την ε, παρουσίαση του, πράσινου, του ε, λευκού βιβλίου ε, και θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Καντράου για τη σημασία των 10 πρώτων ετών, των όσων δηλαδή πρέπει να κάνουμε σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα θέλουμε να πετύχουμε Έπειτα για το χειρισμό της ζήτηση ε, ε, που αναφέρεται στο Λευκό Βιβλίο για, την Κομισιόν, αλλά δεν ε, αναφέρεται από την άλλη πλευρά κανένα μέσο ή κανένα στόχος μετρήσιμος. Επίσης, να εκφράσω τη λύπη μου που δεν ασχολείται το Λευκό Βιβλίο με μια ενδιαφέρουσα δυνατότητα, να εντοπίσουμε δηλαδή σε ποιο βαθμό ποια, μια πιο ευφυής κινητικότητα θα μπορούσε να δημιουργήσει επασχόληση και όχι να οδηγήσει σε απώλεια απασχόλησης ή ανάπτυξης. Δεν είναι υποχρεωτικό η κινητικότητα να οδηγήσει σε λιγότερε θέσει απασχόληση. Αντίθετα, αν βελτιώναμε, αν χρησιμοποιούσαμε την ε, κοινή χρήση αυτοκινήτων, ε, τη χρήση των ε, κοινών μέσων μαζική μεταφορά κτλ., θα οδηγούσαν σε βελτίωση. Δηλαδή οι μεταφορές δεν σημαίνει ότι θα κάνει ο καθένας μόνος του ό,τι μπορεί να κάνει, δηλαδή να είναι ένα self-service, αλλά αντίθετα να χρησιμοποιηθούν διάφορα μέσα για μετακίνηση και μέσα στα αστικά κέντρα με βελτιστοποίηση των μεταφορών. Όλα αυτά θα επέτρεπαν όπως έγινε και στην ενέργεια, να έχουμε μέσω της ε, ε, καλύτερης, πιο οργανωμένης κινητικότητας, να έχουμε μια κινητικότητα που θα οδηγήσει σε περισσότερες θέσεις απασχόλησης, και καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτή η πτυχή λείπει από το Λευκό Βιβλίο και θα πρέπει να εμείς να το επεξεργαστούμε στην εκθεσή μας, ώστε να καταστεί πιο ισχυρή και να έχουμε στόχους πιο ε, βράχοι πρόθεσμους, όχι μόνο με 30 χρόνια. Κύριε Τικάου. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σας καλέσω να σκεφτούμε το λευκό βιβλίο του 2001 που ίσχυε μέχρι το 2010 και να κάνουμε και έναν απολογισμό, να δούμε δηλαδή τι υλοποιήθηκε, τι, ποιοι ήταν οι στόχοι που δεν επιτεύθηκαν. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις εκρήξεις ε, των ηφαιστείων αλλά και τα χιόνια που επηρέασαν τον τομέα των μεταφορών, όχι μόνο των εναέριων μεταφορών. Το, το λευκό βιβλίο μας προτείνει να σκεφτούμε μακροπρόθεσμα μέχρι το 2050, αλλά πιστεύω πως το Λευκό Βιβλίο θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική ε, ε, δομή των ευρωπαϊκών δικτύων, αλλά και ε, να μιλήσει για τη χρηματοδότηση αυτών των δύο ευρωπαϊκών δικτύων. Η διαλειτουργικότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να έχουμε ένα αποτελεσματικό ε, σιδηροδρομικό δίκτυο γιατί η επιφάνεια της Ευρώπης είναι σχετικά μικρή αλλά, με πολύ πυκνο, αλλά είναι πολύ πυκνοκατοικημένη. Να έχουμε λοιπόν αποτελεσματικό σύστημα σιδηροδρομικό θα πρέπει να δούμε και ένα ολοκληρωμένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για τους σιδηροδρόμους. Όσον αφορά τώρα τις οδικές μεταφορές, νομίζω πως θα πρέπει να υπάρξει ισορροπημένη ανάπτυξη στα νέα κρατημέλη, γιατί εκεί οι, οδικοί, οι οδικές υποδομές δεν είναι τόσο αναπτυγμένες όσο στα παλιά κρατημέλη και μέσα στο πλαίσιο το πολιτέ, το δημοσιονομικό πολιτέ πλαίσιο θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτό το ζήτημα και να χρηματοδοτήσουμε τις δομές οδικών μεταφορών στα νέα κράτη-μέλη. Ε, βεβαίως ε, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να αναπτυχθούν τα ΕΦΗ e, συστήματα μεταφορών και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να φτιάξουν εθνικά συστήματα για να επιτευχθεί ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών. Και γι' αυτό είναι σημαντική και, και οι ευρωπαϊκοί κανόνε. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, δεν έχουμε επαρκή χρηματοδότηση και άρα θα χρειαστεί να βρούμε μέσα και πόρου επιπλέον για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών. Τώρα θα ήθελα να τονίσω τους ε, πολίτες ε, που χρησιμοποιούν τα συστήματα μεταφορών αλλά και τους εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών. Θα πρέπει να σκεφτούμε τις συνθήκες εργασίας τους. Για τα άτομα με ειδικέ ανάγκε, για παράδειγμα. Πρόεδρε, ποιο θα είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα αυτά, γιατί θα έχουμε αυτή την έκθεση. Ο κύριο Γκρό ε, είναι πολύ καλό συζητητή, έχει μεγάλη πείρα, το ξέρουμε όλοι αλλά θα υπάρξει αυτό το ψήφισμα που σύμφωνα με τη συνθήκη της Νίκαιας και της Λισαβόνας θα μπορούσε να μας επιτρέψει να απαιτήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα χρόνο μετά από την υιοθέτηση του ψηφίσματος να μας προτείνει νομοθετικές προτάσεις. Μέσα στο πλαίσιο των διοργανικών σχέσεων λοιπόν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να είναι μόνο μια πολιτική δήλωση, στερημένη δράση, αλλά θα πρέπει να ακολουθηθεί από συγκεκριμένε ενέργειε. Ποιε θα είναι λοιπόν οι νομοθετικέ πρωτοβουλίε που θα μπορούσαμε να πετήσουμε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίση το Ελευκό Βιβλίο αντικατοπτρίζει το πρόγραμμα εργασία τη Κομισιόν για την περίοδο 2011-2012. Ο κ. Αλκαντράου έλεγε πω δυστυχώ οι περισσότερε δράσει είναι ε, προγραμματισμένε για το δεύτερο ήμιση του χρόνου, αλλά εμεί θα θέλαμε να γνωρίζουμε Ποιε είναι οι συγκεκριμένες δράσεις για την επόμενη περίοδο. Ευχαριστώ. Ο κύριο Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχοντα ε, διαβάσει τα έγγραφα, έχω δύο, ε, έχω δύο απόψεις. Ε, πρώτον, ε, το ε, έγγραφο αυτό θα, ε, θα λήξει κάποια στιγμή και θα χρειαστούμε κάποιο καινούριο. Μπορεί λοιπόν κανεί να πει ότι επί της αρχής μπορούμε να υιοθετήσουμε την Λευκή Βίβλο αυτή. Ε, έχουμε καταλήξει κάπου, αλλά κάτι λείπει. Εάν κοιτάξουμε την προοπτική 20 συν 20, δηλαδή το 2050, Ποιοι θα είμαστε σε 20 ή 40 χρόνια, ποια θα είναι τα επίπεδα ΑΕΠ και τι θα ισχύει όσον αφορά την ε, αποσύνδεση ή τη σύνδεση. Θα, διπλασιάσουμε τις μεταφορές μας μέχρι τότε. Θα γίνουν σίγουρα ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές μέχρι τότε. θα πρέπει να εξετάσουμε και τι δυναμικό θα χρειαζόμαστε όσον αφορά τα συστήματα μεταφορών. Ε, θα έχουμε ποιοτική ή ποσοτική ανάπτυξη και αν ε, θα είναι ε, ποιοτική πώς θα την πετύχουμε και πάλι θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα προχωρήσουμε βήμα προς βήμα ότι θα ενισχύσουμε την πρόταση της Κομισιόν με τη συνεργασία των κρατών μελών ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ε, σε τι βαθμό χρησιμοποιούμε εδώ την ευρωπαϊκή μέθοδο. Θα έχουμε ένα σύστημα ε, για όλη την Ήπειρο ε, για τις αερομεταφορές ή για τους αυτοκινητοδρόμους. Δεν βλέπω να υπάρχει εδώ αυτή, αυτό το στοιχείο που να καλύπτει το σύνολο της Ήπειρου της Ευρώπης το όραμά μας θα πρέπει να το εξετάσουμε και ε, σε σχέση με το ε, περιβάλλον. Θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με το παγκόσμιο περιβάλλον και πάνω απ' όλα οι μεταφορές ε, θα αυξήσουν τον ανταγωνισμό. Και μία ερώτηση ακόμα. Πριν 40-50 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι χώρες δημιούργησαν μεγάλα ε, έργα υποδομής, ενώ σήμερα δυσκολευόμαστε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τι ε, πάει στραβά στο ευρωπαϊκό σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λίγα λόγια και από μένα, αν μου επιτρέπετε. Πάντα θεωρώ ότι είναι εύκολο να είναι κανείς αρνητικός απέναντι σε μια τόσο μεγάλη έκθεση ή ένα τόσο μεγάλο κείμενο όσο αυτό. Σίγουρα είναι ε, ενδιαφέρον να ακούμε τις ε, διάφορες απόψεις. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπερβολικά ριζοσπαστικό το κείμενο, άλλοι θεωρούν ότι δεν ε, κάνει αρκετά. Προσλέπω λοιπόν να ακούσω τον κύριο Γκρός να κάνει τον Σολομόντα και να προσπαθήσει να βρει μια μέση οδό όσον αφορά το πόσο ριζική είναι τελικά η Λευκή Βίβλος. Εγώ την εξέτασα και διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά δεν βλέπω πουθενά στην έκθεση να λέει ότι θα πρέπει να απαγορεύσουμε τα αυτοκίνητα. Θα πρέπει λοιπόν καταρχήν να ε, εξαλείψουμε αυτόν τον μύθο. Καταρχήν δεν μιλάει για τέτοιο πράγμα. Λέει ότι θα πρέπει να έχουμε ε, κέντρα πόλεων απειλαγμένα από οχήματα ορυκτών καυσίμων. Πουθενά όμως δεν λέει ότι θα πρέπει να απαγορεύσουμε γενικά τα αυτοκίνητα. Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, Όσον αφορά το να αφήσουμε την αγορά να τα αποφασίζει όλα, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη και ρόλος για την αγορά, αλλά η αγορά δεν είναι κάποιος θεός. Το να αφήσουμε την αγορά να αποφασίσει τα πάντα, κατά τη γνώμη μου, είναι συνταγή για την καταστροφή. Πρέπει να υπάρχει κάποια ισορροπία και γι' αυτό δεν μπορώ να ακολουθήσω το επιχείρημα ότι ε, θα κάνουμε ό,τι αποφασίσει τελικά η αγορά. Ε, στον ε, χρηματοπιστωτικό τομέα η αγορά αποφάσισε κάτι το οποίο ακόμα μας στοιχειώνει. Και επικροτώ τη συμπερίληψη του κοινωνικού στοιχείου. Και υπάρχει εδώ μια πρόκληση. κυρία Φώστερ ε, εγώ αμφισβητώ αυτό που είπατε ότι θα πρέπει να ασχοληθεί η Επιτροπή ε, Απασχόλησης. Μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό διότι εξετάζουμε τον τομέα και κοιτάμε το πώς... Ε, το τι μεταχείριση έχουν οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές στον τομέα των μεταφορών και αυτό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τομέα των μεταφορών και πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τα πρότυπα του τομέα. Εμείς όσοι υπεύθυνοι για τις μεταφορές θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να λέμε αν είναι ε, καλά τα στοιχεία αυτά κακά ή ε, αδιάφορα. Δεν είμαι διατεθειμένος να αφήσω οτιδήποτε έχει σχέση με την απασχόληση στην Επιτροπή Απασχόλησης και το ίδιο ισχύει για τα περιβαλλοντικά θέματα και την ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ε, όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών, εγώ δεν έχω χορτάσει με το θέμα αυτό. Εγώ είμαι ικανοποιημένο με τα δικαιώματα των επιβατών που έχουμε, αλλά μερικέ φορέ ε, πρέπει να. Ε, αναρωτιόμαστε γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν απαραίτητο να νομοθετήσουμε όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. μήπω επειδή η αγορά δεν φρόντιζε επαρκώς τον καταναλωτή και ε, επειδή ε, είχαν κακή μεταχείριση οι επιβάτες ε, και πάλι εναπόκειται σε εμά να νομοθετήσουμε, να φροντίσουμε να προστατεύονται οι επιβάτες από τις υπερβολές. Στα πλαίσια της Λευκής Βίβλου θέλουμε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό όραμα και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες διστάμενες απόψεις. Ξέρουμε ότι ε, τα κράτη-μέλη ε, έχουν ε, οπισθοχωρήσει όσον αφορά το θέμα των εθνικών συνόρων. Εγώ θέλω να υπερασπιστώ την ε, ε, ε, την ευρωπαϊκή διάσταση εδώ και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που περιλαμβάνει και ευθύνη απέναντι όχι μόνο στους επιβάτες και στους καταναλωτές αλλά απέναντι και στις επιχειρήσεις. Ε, στόχος είναι να βρούμε μια ισορροπία εκεί. Είμαι αισιόδοξο λοιπόν ότι με τον εισηγητή μας μπορούμε ως κοινοβούλιο να προχωρήσουμε, να συνεργαστούμε με την Κομισιόν καθορίζοντας τα στοιχεία του οράματος για το 2050. Συμφωνώ ότι θέλουμε κάποια περισσότερα ε, ενδιάμεσα βήματα. Ε, ξέρω ότι είναι πολύ απίθανο να είμαστε εδώ το 2050. Θα ήθελα όμως ε, να καθορίσουμε κάποιους στόχους για το 2020, το 2030 και το 2050. Κάθε τόσο νομίζω πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο πιο θετικά. Κύριε Γκρός, θέλετε να επανέλθετε. Ναι, σας ευχαριστώ. Δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια πράγματα, απλώς ε, θα ήθελα πολύ σύντομα να πω ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή εδώ πιστεύω στη δουλειά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χάρη στην έκθεση αυτή. Το ακούσαμε σε τελευταία ανάλυση και από άλλους ε, συναδέλφους ότι ε, θα πρέπει να γίνει μια βασική επιλογή για το εάν η ελεύθερη αγορά μπορεί να δώσει τις απαντήσει σε όλα τα προβλήματα από μόνη της ή εάν οι εθνικές αγορές μπορούν να επιλύσουν όλα τα προβλήματα. Πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε ε, θαραλέοι και να αντιμετωπίσουμε ορισμένε και λαϊκιστικού χαρακτήρα μάλιστα δηλώσει, οι οποίε λένε ότι μπορεί το κάθε κράτο μέλο να ορίσει μόνο του τι θέλει, χωρί ε, να λαμβάνει υπόψη ότι ισχύει στα γειτονικά κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι και από την οικονομία και τη βιομηχανία ξεκάθαρα απευθύνεται το μήνυμα δώστε μας πιο ενιαίους κανόνες ε, Δώστε μας συνθήκες εργασίες, εργασίας όπου δεν μπορεί κανείς να ανησυχεί ότι μπορεί στο γειτονικό κράτος να ισχύσει κάτι διαφορετικό που θα οδηγεί σε κοινωνικό ή εργασιακό dumping ή σε συνθήκες διαφορετικές απασχόλησης. Άρα λοιπόν, όταν μπορούμε να έχουμε κάποια ε, λύση εθνική ικανοποιητική τότε δεν χρειάζεται να παρεμβαίνει ε- η Ευρώπη. Αλλά όταν βλέπουμε ότι οι εθνικές ρυθμίσεις αποτελούν πρόσκομα μάλλον στην εξέλιξη, τότε θα πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα όραμα για τις μεταφορές που θα διευκολύνει και τη ζωή του πολίτη και την λειτουργία της οικονομίας. Απλώς αυτό θα πρέπει να το καταστήσουμε λίγο πιο σαφές, ενδεχομένως και σε επίπεδο της Επιτροπής μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη τα, το 2050 ως ορίζοντα, αλλά ε, χωρίς να λησμονούμε ότι πρέπει πρώτα να δώσουμε κάτι πιο σύντομο ως προοπτική με συγκεκριμένα μέτρα. Επίσης θα ήθελα να πω ότι η πολιτική είναι πολιτική απόφαση για το πού θα πάνε τα χρήματα που είναι διαθέσιμα. Σε κάθε κράτος χρήματα εκτός από ίσως ένα-δύο, μια-δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, χρήματα υπάρχουν. Ε, και πάλι και στα άλλα κράτη θα, υπάρξουν κάποια στιγμή. Εν πάση όμως πρέπει να γίνει η επιλογή το πού θα πάνε τα χρήματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν ορίσει έναν κατάλογο 300 προτεραιοτήτων για τι μεταφορέ, δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Όμω έχουμε το θάρρο, να επικεντρωθούμε σε 15 συγκεκριμένα σχέδια, να πούμε ότι ε, εστιάζουμε τη χρηματοδότησή μα με βάση το ποσοστό 10, 15, 20, 30, αλλά και εφόσον και με προπόθεση τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα από πλευρά του να φέρουν μέρο του οικονομικού αυτού βάρους, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Αν δεν το πράξουμε, θα έχουμε αποτύχει. Και η χρηματοδότηση, όπως είπα, είναι βαθιά μου πεποίθηση ζήτημα πολιτικής βούλησης. Εάν δεν θέλουμε να επενδύσουμε στις υποδομές, δεν χρειάζεται μετά να διαμαρτυρόμαστε αν δεν έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε σε ορισμένους τομείς στη συνέχεια στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ τις πολιτικές ομάδες για την πολύ καλή συνεργασία στην οποία προσβλέπω. Μπορεί να μην έχουμε πάντοτε τις ίδιες επόψεις, αλλά είμαι βεβαίως ότι θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία και θα καταλήξουμε σε καλές προτάσεις. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι είναι απέτηση γενική να διατυπωθούν σαφείς ε, προτάσεις και ορόσημα για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ουγκρό. Το σχέδιο εκθέσεως προβλέπεται για το Σεπτέμβριο. Η εξέταση των τροπολογιών προβλέπεται να γίνει στις 10 και 11 Οκτωβρίου με ψηφοφορία στην Επιτροπή των Μεταφορών στα τέλη του μηνός Νοεμβρίου. Προς το παρόν αυτό προβλέπεται και ελπίζω να μην έχετε αντίρρηση κύριε Γκρός. Σας ευχαριστώ. Το επόμενο θέμα στην εμερησία διάταξη είναι το παλαιό και γνωστό θέμα του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Εξέταση των τροπολογιών με εισηγήτρια την κυρία Σερρακιάνη που έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. πριν ξεκινήσεις ε, Δέμπορα, παρακαλώ μπορείτε ήδη να ζητήσετε το λόγο ώστε να δω πόσο χρόνο έχουμε και να μοιράσω το χρόνο δίκαια. Συγγνώμη, δεν να συνέχισε. Ναι, ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους εισηγητές, τους Σκιώδης, με τους οποίους ε, συναντήθηκα αρκετές φορές. Ε, θα συνεχίσω να τους ε, συναντώ συχνά όπως να ευχαριστήσω και τους βουλευτές της Επιτροπής Μεταφορών που με βοήθησαν στην σύνταξη αυτής της πρώτης πρότασης. Ε, μόνο 597 τροπολογίες πήρα. Για να είμαι λοιπόν πιο σαφή στην παρουσίασή μου, προτίμησα να περιοριστώ σε κάποια και να τις χωρίσω σε βασικά επιχειρήματα. Πρώτο, επιχείρημα, πρώτο θέμα είναι το θέμα του ρυθμιστή, δεύτερο είναι η ανεξαρτησία του διαχειριστή των υποδομών, έπειτα ο τομέας το συνδυνομικός ή το άνοιγμα της αγοράς και έπειτα οι βασικές υπηρεσίες. Φυσικά δεν είναι ε, ε, πλήρης αυτός ο κατάλογος, αλλά είναι τα πιο σημαντικά ε, θέματα. Όσον αφορά τον ε, ρυθμιστή, υπήρξαν τροπολογίες για το άρθρο 55 που αφορά την οργάνωση του ρυθμιστή. Ορισμένες από αυτές τις τροπολογίες τις είμαι σύμφωνη και εγώ γιατί είναι τροπολογίες που προσπαθούν να ενισχύσουν, να εγγυηθούν την οργανωτική, τις οργανωτικές δυνατότητες του ρυθμιστή, καθώς και να εγγυηθούν τις δυνατότητες του ρυθμιστή αυτού να όχι. Διακόπτη. Η ομιλήτρια... Α, δεν είναι δικό μου το πρόβλημα. Να εγγυηθεί λοιπόν την οργανωτική δυνατότητα του ρυθμιστή καθώς και να προβλέψει το ότι θα έχει τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες ε, πιο συγκεκριμένα που ενισχύουν όπως αυτή του κυρίου μπαχ που ενισχύουν την υποχρέωση διαφάνειας για τους φορείς που λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο του ρυθμιστικού φορέου. Πολλές τροπολογίες επίσης συμπεριλαμβάνουν την αρχική μου πρόταση σε σχέση με τον διορισμό ή την επικύρωση του Εθνικού Κοινοβουλίου για τον ρυθμιστικό φορέα. Υπήρξαν τροπολογίες και για τα άρθρα 56 και 56α που αφορούν τις εξουσίες της αρμοδιότητας του ρυθμιστικού φορέα. Ας πούμε, ο κύριος Τρεμόζα ζητά να θεσπιστεί ε, μια διορία για την υιοθέτηση της απόφασης από πλευράς του ρυθμιστικού φορέα. Υπάρχουν διάφορες υποδείξεις. Ο κύριος Τρεμόζα επέδειξε δύο εβδομάδες, ε, ε, οι άλλοι πρότειναν 20 εργάσιμες μέρες. Εν πάση περιπτώσει ζητήθηκε και η δυνατότητα από πλευρά ε, εφετείου, μάλλον κάτι σαν εφετείο, μετά από 20 ε, εργάσιμες ημέρες, ο κύριος Κούν επαναφέρει την αρχική πρόοδο, του, την αρχική μάλλον διορία του ενός μήνα. Ε, υπάρχουν διάφορες τροπολογίες που υποβλήθηκαν και για τις εξουσίες που μπορεί να έχει ο ρυθμιστικός φορέας, αλλά και για την ίδια τη δυνατότητα, δηλαδή να προβλέπονται και κυρώσεις. Ορισμένες τροπολογίες προσπαθούν να καθορίσουν συγκεκριμένες κυρώσεις και πρόστιμα και ακυρώνουν το ρόλο του επόπτιο για τον ίδιο τον αριθμιστικό φορέα για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους ετούντες και τους διαχειριστές των υποδομών σε σχέση με το επίπεδο δικαιώματος χρήσης της υποδομής. Για το άρθρο 57 που αφορά την συνεργασία ανάμεσα στους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και εδώ υποβλήθηκαν διάφορες τροπολογίες που εν έχουν συμπεριλάβει και τη δική μου αρχική ιδέα να υπάρξει ένα επίσημο δίκτυο υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η τροπολογία 628 για παράδειγμα του κυρίου Κόζα έχει στόχο τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για τις ε, ε, για τις ε, καταγγελίες. Ε, επίσης γίνεται πρόταση για την ένταξη αυτής της αρχής στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Υπάρχουν άλλες τροπολογίες σε σχέση με το δίκτυο των ρυθμιστών, της κυρίας Βλαστό και άλλων που θα υποχρέωναν το δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων να αναλαμβάνουν την επίλυση διαφορών που αφορούν περισσότερα από ένα κράτος. Ε, υπευλήθησαν και τροπολογίες του κυρίου Καντσάν και Φιντάντσα που ενισχύουν το ρόλο της Κομισιόν σε σχέση με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές. Υπάρχουν και παρεμβάσεις τις οποίες συμμερίζομαι που αφορούν τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα. Τροπολογίες, ε, μάλλον έτοιμα το οποίο υπήρχε και στο πρώτο μου σχέδιο έκθεσης. Άλλες τροπολογίες ενισχύουν το ρόλο των αριθμιστικών φορέων για το, την χάραξη των διεθνών διαδρομών, ενώ άλλες τροπολογίες αρνούνται κάθε λειτουργία που μπορεί να έχει ένας αριθμιστικός φορέας ως παρατηρητής σε σχέση με τις συνεδριάσεις που γίνονται από τους διαχειριστές των υποδομών. Υπάρχει δηλαδή διαφορετική ιδέα σε σχέση με το ποιε θα είναι οι αρμοδιότητες που θα έχει ο Εθνικός Αριθμιστικός Φορέας και ως προς αυτό και σε σχέση με τις εξουσίες της Επιτροπής. Όπως έχω ήδη πει, θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω ένα κείμενο το οποίο να περιλαμβάνει μια ενίσχυση της θέσης ε, του ρυθμιστικού φορέα καθώς και τη δυνατότητα ενός δικτύου ρυθμιστών, τη δυνατότητα για μια πιο στενή συνεργασία. Άλλο σημαντικό σημείο που αφορά την ανεξαρτησία των διαχειριστών ε, των υποδομών. Εδώ χρειάστηκε εν μέρει να αλλάξω τη θέση μου για να προσπαθήσω να βρω μια πολιτική συμφωνία, γιατί πιστεύω πως είναι σημαντικό να σταλεί ένα πολιτικό μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση και θα ήθελα πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή Μεταφορών να εκφραστεί πολύ πιο ε, έντονα για αυτό το θέμα και γι' αυτό υποβλήθηκαν και τροπολογίες που εν μέρη άλλαξαν την αρχική δομή του πρώτου σχέδιου έκθεσης ε, τροπολογίες τις οποίες εν μέρη υπέβαλα εγώ και, στις, και τις έχει συνυπογράψει και ο κύριος Κούρνα. Στόχο έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια για την ε, χωριστή λογοδοσία των διαχειριστών των υποδομών. Ξεκαθαρίζουν τις αρμοδιότητε των διαχειριστών των υποδομών από τη μια πλευρά και του ε, ε, φορέα του δικτύου από την άλλη πλευρά. Επι, για παράδειγμα, υπάρχει δυνατότητα διατήρησης του holding, του ομίλου, όπως υπάρχει σε ορισμένες χώρες. Στα όσα θύμισα έτσι γενικά, υποβλήθηκαν δύο ομάδες τροπολογιών. Από τη μια πλευρά έχουμε αυτές που θέλουν να τονίσουν τις χωριστούς ε, λογαριασμούς και από την άλλη πλευρά μια ομάδα τροπολογιών που στόχο έχουν να αποδυναμώσουν το αίτημα των χωριστών, ε, της χωριστής λογοδοσίας και της ανεξαρτησίας του, της υποδομής. Όσον αφορά τις πρώτες, να θυμίσω αυτούς που θέλουν να ενισχύσουν την ε, χωριστή τη χωριστή λογοδοσία, η κυρία Γιάλα ζητά να απαγορευτεί η μεταφορά κονδυλίων από, ανάμεσα στι διάφορε ε, Από την άλλη πλευρά, Καντζάν και Φιντάντζα ζητούν να υποδειχθούν ποια είναι τα κριτήρια αναξαρτησίας θα, θα πρέπει να τηρεί ο διαχειριστής της υποδομής όταν πρόκειται για βασικέ λειτουργίε και ο κύριο Τρεμόζα ζητά την απαγόρευση τη μεταφορά προσωπικού management τη υποδομή για μια τριετή περίοδο. Όσον αφορά αντίθετα τις τροπολογίες που στόχο έχουν να αποδυναμώσουν αυτήν την, την, την ανεξαρτησία έχουν υποβληθεί διάφορες σχετικέ τροπολογίε από τον κύριο Βίλς, για παράδειγμα, που ζητά εξαίρεση στην απαγόρευση της μεταφοράς δημοσίων κονδυλίων σε περίπτωση υπηρεσιών κοινή ωφέλεια. Ε, μια τροπολογία του κυρίου Μπάκα που αφορά την μέθοδο διαρθωτικού διαχωρισμού που θα πρέπει να επιτρέψουν να διατηρηθεί ο ανταγωνισμό και οι επενδύσει. Τρίτο θέμα, ε, εξίσου σημαντικό, είναι το θέμα της χρηματοδότησης του σιδηροδρομικού τομέα που αφορά τα άρθρα 8 και 9 και εδώ υπήρξαν ε, πολλοί άρθμες τροπολογίες. Σημερίζομαι τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν από τους κυρίους Ζήλε και Γκρός, με τις οποίες θα ζητούν τα κράτη-μέλη να καλύπτουν ε, τις υπόλοιπες ε, δημοσιονομικές ανάγκες των διαχειριστών των δικτύων για να εγγυηθούν την ανάπτυξη της ίδιας της υποδομής. Υποβλήθηκαν επίσης τροπολογίες που ενισχύουν τη διαδικασία διαβούλευσης με τα συνδικάτα και τις τοπικές αρχές και άλλες τροπολογίες ζητούν να ακυρωθεί η μη δεσμευτική γνωμοδότηση του φορέα για το business plan, ενώ άλλες ε, κατά κάποιο τρόπο ζητούν να αποδυναμώσουν την υποχρέωση εξισορρόπησης ε, των ε, λογαριασμών ανάμεσα στους διαχειριστές των υποδομών. Τροπολογίες υποβλήθηκαν επίσης από πολλούς συναδέλφους. Τώρα εγώ προσωπικά δεν θα ήμουν αντίθετη στο άνοιγμα της αγοράς, αλλά φυσικά θα περιοριστώ στην απόφαση της πλειοψηφίας. Τη επιτροπή Μεταφορών σε σχέση με το κατά πόσο θα λάβουμε υπόψη τη δυνατότητα ένταξης στο σχήμα της αναδιατύπωσης και τα αιτήματα τα οποία σχετίζονται με το άνοιγμα τη αγορά. Όπως σας έλεγα υπάρχουν διάφορες τροπολογίες, ε, κατά βάση αυτές υποβλήθηκαν από τον κύριο Τρεμόζα, Ρικέ, Καντζάν και Φιντάντζα, που εισάγουν αυτό το αίτημα ανοίγματο του εθνικού ανοίγματο της ε, μεταφοράς επιβατών. Υπάρχει μια τροπολογία Φιντάντσα Καντσάν που ζητά το άνοιγμα της αγοράς και μάλιστα με μια ρήτρα αμοιβαιότητα σε σχέση με τις κλειστέ αγορές, ενώ και σχέση με αυτό το άνοιγμα υπάρχουν φυσικά αντίθετες απόψεις που θέλουν να διατηρήσουν κάποιες εξαιρέσεις όσον αφορά τις ε, υπηρεσίες κοινή ωφέλεια. Για την άλλη ομάδα τροπολογιών, τις οποίες ε, συνδύασα στις βασικές υπηρεσίες που αφορούν ε, δηλαδή το άρθρο 13, να θυμίσω μόνο ο τίτλους κάποιων τροπολογιών. Για παράδειγμα, το άρθρο 13... Είναι πολλές τροπολογίες που υποβλήθηκαν ε, στην υποπαράγραφο 1 του άρθρου 13 που αφορά τις βασικές υπηρεσίες. Ε, υπάρχει ένα αίτημα για διάφορες μάλλον τροπολογίες που προτείνουν την ακύρωση αυτής της υποπαραγράφου που υποχρεώνει σε ένα μίνι, μίνι αποδέσμευση για τους φορείς και προτείνουν ότι κατασταθούν ορισμένε πιο ελαφριέ διατάξει όπως οι χωριστοί λογαριασμοί ή τα αιτήματα για διαφάνεια. Και εδώ και για αυτή την ομάδα υπάρχουν πολλοί άριθμες τροπολογίες Ο κύριο Τρεμόζα, σε σχέση με την υποπαράγραφο 4, θα ήθελε ο ρυθμιστή να έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει εναλλακτικέ λύσει όταν λείπει η δυνατότητα ανταπόκριση σε όλα τα αιτήματα, ενώ άλλοι, όπω για παράδειγμα η ομάδα των Πρασίνων, ζητούν να ακυρωθεί οποιαδήποτε επαναφορά στο ρόλο του ρυθμιστή στην επίλυση ε, διαφορών. Σε σχέση με αυτό το άρθρο, όπως σα είπα, είναι πολύ άριθμε οι τροπολογίε. Υπάρχουν και άλλα ε, θέματα τα οποία εδώ δεν ανέφερα, δηλαδή δεν τα έχω εντάξει στις πέντε πιο σημαντικές ομάδες τροπολογιών, που όμως είναι η παρακολούθηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, δάσου 15, και εδώ υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί με βάση τη συνεργασία για, μεταξύ διαφόρων φορέων, δηλαδή συνδικάτων, κοινοβουλίων, διαφόρων φορέων, ώστε να ε, συμπεριληφθούν νέα στοιχεία στον κατάλογο των αγορών. Υπάρχουν και τροπολογίες που σχετίζονται με το κόστος. Τα άρθρα 29 με 37 αφορούν το κόστος και εδώ υπάρχουν τροπολογίες που ζητούν για παράδειγμα την κατάργηση από πλευρά του ρυθμιστικού φορέα για την επαλήθευση των εσόδων τροπολογίες 501 και 504, ενώ υπάρχουν άλλες τροπολογίες αντίθετα που θέλουν να ενισχύσουν τον έλεγχο του ρυθμιστικού φορέα, για παράδειγμα, για την αναθεώρηση των ε, συμβάσεων, για το θόρυβο. Ο, η ομάδα των Πρασίνων προτείνουν να καταστεί υποχρεωτικό, αλλά θα πρέπει να παραμείνει ουδέτερο το θέμα του κόστου σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν για το θόρυβο για τον οδικό τομέα. Υπάρχουν και προτάσεις τροπολογίας που ζητούν να συνδεθεί το θέμα του κόστους που προβλέπεται στην αναθεωρημένη οδηγία με τα όσα θα συμβούν σε άλλους τομείς μεταξύ των οποίων και η οδική μεταφορά εμπορευμάτων. Και άλλες τροπολογίες αφορούν το τμήμα για την καινοτομία, για τα δίκτυα MS, τα συστήματα τα οποία, για τα οποία δίνονται κίνητρα μέσω της αναδιατύπωσης ώστε να ενταχθούν κάπως σε αυτό τον ενιαίο αγορά. Έπειτα και θυμίζω δύο ακόμα ζητήματα που δεν είναι όμως ε, περιφερειακά και αφορούν τον ορισμό των υποδομών που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1 και εδώ υπάρχουν τροπολογίες και έπειτα το ζήτημα που σχετίζεται με τις πράξεις κατεξουσιοδότηση σε σχέση με αυτές δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο αίτημα του κατά πόσο θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πράξεις, ναι ή όχι, αλλά ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε ποιες ποιο θα ήταν το περιεχόμενο που καλύπτεται από άρθρα τα οποία ήδη συμπεριλαμβάνονται στις πράκτικα της εξουσιοδότηση ή στην εφαρμογή όπως αποκαλείται ε, ώστε να μην υπάρξει αντίθεση σε σχέση με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Σε σχέση με τα όσα έγιναν για την αναβολή της ψηφοφορίας που προβλεπόταν για τον Ιούλιο και που αντίθετα αναβλήθηκε, όσο με αφορά εγώ θα συνεχίσω τις επαφές μου με τους σκιώδεις εισηγητές. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε δηλαδή πάνω στο κείμενο, θα προτιμούσα να μην είχε υπάρξει αναβολή, γιατί θα ήταν ένα σημαντικό μήνυμα να δείξουμε ότι σε σχέση με το σιδηροδρομικό σύστημα δίνουμε προσοχή και σε σχέση με τις γραμμές που αναφερθήκαμε πριν σχολιάζοντας ε, το λευκό βιβλίο ότι, υπάρχει, ότι δίνεται προσοχή από πλευρά τη Κομισιόν στο σιδηροδρομικό τομέα. Ωστόσο, ζητήθηκε αναβολή για να εξεταστούν καλύτερε συμβαστικέ προτάσει. Άρα λοιπόν πάμε για μετά το καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Thank you very much. Just... Ευχαριστώ πολύ για να ενημερώσω την εισηγήτρια αλλά και τους συναδέλφους. Προβλέπω μια περαιτέρω συζήτηση τον Αύγουστο στη συνεδρίασή μας, όπου ελπίζω ότι με τις διαπραγματεύσεις που θα έχουν γίνει θα έχουμε την ευκαιρία να συστήσουμε περισσότερο επί, τη, επί των συμβαστικών τροπολογιών παρά των, επί των επιμέρους. 30-31 Αυγούστου που έχουμε τη συνεδρίαση. Πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε εξασφαλίσει τις συμβαστικές προτάσεις και όπως είπατε και εσείς, ψηφοφορία τον, Αύγου, τον Οκτώβριο και για την Ολομέλεια τον Νοέμβριο. Άρα ας προσπαθήσουμε στο χρόνο που έχουμε στη, στη διάθεσή μας εντωμεταξύ να ε, βρούμε συμβαστικέ τροπολογίε. Έχω αρκετού ομιλητέ όπω φαντάζεστε. Οι σκιώδει θα λάβουν από 6 λεπτά, οι λοιποί από 4. Πρώτο σκιώδη είναι ο κύριο Κούν. 6 λεπτά όπω είπα. Οι σκιώδει ηγητέ και από τέσσερα τα λοιπά μέλη τη Επιτροπή. Έχω 14 με 15 συναδέλφου που να λόγο. Κύριο Κούν. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ και την εισηγήτρια, την κυρία Σαρακιάνη, για την δουλειά που έχει αναλάβει. 736 τροπολογίες προφανώς καθιστούν το έργο της αρκετά δύσκολο όπως θα προσδιορίσει τις προτεραιότητες και και καλό θα είναι να μην χρειάζεται να δουλεύει υπό πίεση χρόνου. Νια χρόνια δεν μπόρεσε η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη να ρυθμίσει το θέμα αυτό και τώρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να διαφετήσουμε την υπόθεση των συντηροδρομών ε, μέσα σε διαδικασίες ε, ε, επιταχυμένες. Και πρέπει να προσδορίσουμε προτεραιότητες, πιστεύω. Μια πρώτη προτεραιότητα στην οποία συμφωνούμε είναι ότι θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να έχει μια ρυθμιστική αρχή, να θεσπίσει ρυθμιστική αρχή η οποία θα ακολουθεί τις ίδιες δομές, οι ανάλογες δομές με τον λοιπόν θα έχει μια πρικοδότηση οικονομική, υλική, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό ικανή θα έχει αρμοδιότητες για την ε, διεκπαιρέωση όλων των θεμάτων των σχετικών με τον ανταγωνισμό και πρόσβαση στο δίκτυο, στα δίκτυα παραμένει το κύριο και σοβαρότερο θέμα. Άλλωστε σε αυτό, ε, αυτό προσεγγίζουν οι προσθέρες τροπολογίες. Χρειαζόμαστε συνθήκες ανταγωνισμού ισότιμες, ε, και για την συμμετοχή στα δίκτυα και για την αξιοποίησή τους, αλλά και για την ε, ηλεκτρική ενέργεια, και το ρεύμα που κινείται ε, ε, το σιδηρόδρομο μέσα σε συνθήκες ασφάλειας δικαίου. Έτσι λοιπόν η ρυθμιστική αρχή έχει κύρια, κύριο καθήκον τον, και τον ανταγωνισμό και τη διαχείριση των δικτύων κατά τρόπο ισότιμο και δίκαιο. Και χρηματοδότηση και συμφωνία ως προς τις ε, επιδόσεις ε, μεταξύ κρατών μελών και των διαχειριστικών αρχών των δικτύων τους που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εισηγήτρια αντιπροτείνει ε, περίοδο. Λογική πιστεύω πρόταση και μπορούμε να την, ε, να την προβλέψουμε στη χρηματοδότηση, αλλά αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και τον αντίστοιχο προπολογισμό πλευρά του κράτου μέλου, έτσι ώστε οι υποδομέ που θα προκύψουν και να είναι ικανέ να δώσουν αποτέλεσμα, αλλά και να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά τη διαλειτουργικότητα, ώστε να μην αντιμετωπίζουμε φραγμού και προσκόμματα τεχνολογικού χαρακτήρα. Και δεν θέλω να περάσω επίση το θέμα τη ε, μεταφορά των επιβατών και τη δυνατότητα κάποιο να ξεκινάει φερρυπίν από το Βερολίνο ή τη Βαρσοβία, από τη Βαρσοβία α πούμε μέσω του Βερολίνου με ένα τρένο υψηλής ταχύτητας για να πάει μέχρι το Παρίσι, αλλά ε, να έχει και αντίστοιχα τη δυνατότητα να περάσει από τον σταθμό του τρένου υψηλή ταχύτητα στο κέντρο της πόλης, δεν είναι αυτή το Βερολίνο, είτε είναι το Παρίσι, είτε είναι η Βαρσοβία, με τα κατάλληλα μέσα, ε, σε τροχιά πάλι. Αυτό δεν έχει προβλεφθεί, θα πρέπει να δώσουμε τις λύσεις για το, διαχείριση των υποδομών τώρα. Είμαι ευγνώμων για την, προς την εισηγήτρια. Αρχικά είχε διαγράψει τα άρθρα 6-7 και τώρα βλέπω ότι επαναφέρει ε, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα τα μοντέλα που προβλέπονται ε, να μπορούν να διατηρηθούν και παράλληλα να επιτρέψουν τη λειτουργία το ένα του άλλου χωρίς να παραβλάπτεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η συνύπαρξη τους. Πολλοί είναι οι συνάδελφοι από την ομάδα του ΕΛΚΑ που μου ζητούν να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και να περιγράψουμε τις συνθήκες πλαισίου που θα επιτρέψουν την ικανοποιητική λειτουργία των μοντέλων αυτών θα ήθελα λοιπόν να σημειώσω προς τους συναδέλφους μου, τους οποίους ιδιαίτερα έχουμε συζητήσει αλλά και προς όλους ότι χρειάζονται κόκκινες γραμμές και εγγυήσει ότι δεν θα υποβαθμιστεί το σύστημα σε επίπεδο τέτοιο που ε, δεν θα λειτουργεί ικανοποιητικά. Επίσης και εν προκειμένου έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν για το 2012 σκοπεύει να καταθέσει πρόταση για την αποδέσμευση του unbundling ε, ε, στο σύνολό της γιατί Έχουμε αυτή τη στιγμή ακόμη 22 διαδικασίες επί παραβάση του δικαστήριο που εκκρεμούν ενώπιν του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δηλαδή, μένουν ακόμη ασαφείς οι εξελίξεις και ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να τοποθετηθούμε εμείς σε όλες αυτές τις υποθέσεις, στην, ε, στο μεγάλο θέμα της αποδέσμευσης. Και γι' αυτό θα ήθελα να γνωρίζουμε πώς θα κινηθούμε, ώστε να αποφύγει το Κοινοβούλιο να εμπλακεί σε ένα πλέγμα ε, προβλημάτων αξίας μάλιστα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, γιατί έχουμε να κάνουμε και με τη σιδηροτροχή, έχουμε να κάνουμε με τις ε, σύραγγες, έχουμε να κάνουμε με τον εξοπλισμό των λοιπόν μέσα σε αποφάσεις οι οποίες ενδεχομένως στη συνέχεια να ανατραπούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ή να εξελιχθούν με διαφορετικές αποφάσεις προς διαφορετική κατεύθυνση. Ελπίζω δε και το Συμβούλιο στο ε, εκεί μέλλον να λάβει σαφείς τοποθετήσεις για το θέμα αυτό. Και γι' αυτό πιστεύω και είναι εδώ η δουλειά αυτή ενδιαφέρουσα για όλους. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία και καλές συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ Τρεμόζο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητή Δέμπορα, καλησπέρα. Καταρχήν, ε, επικροτώ την ε, αναβολή της συζήτησης ε, στην Επιτροπή Μεταφορών, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε και να βελτιώσουμε τις τροπολογίες και για να διαβάσουμε την νέα μελέτη του, της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τις βρετανικές εμπειρίες με το unbundling. Για μας, τους φιλελεύθερους, ε, σημαντικό, είναι οι ε, αγορές να είναι ανοιχτές ε, και γι' αυτό προτεραιότητα έχει το ρυθμιστικό πακέτο. Πολλές τροπολογίες συναδέρφων επικεντρώνονται στην σημασία ισχυρών και ανεξάρτητων εθνικών ρυθμιστικών φορέων με επαρκές προσωπικό και πόρους. Ε, θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στην ε, δημιουργία των φορέων αυτών. Οι ε, τροπολογίες μου ζητάνε απόλυτα ανεξάρτητους ρυθμιστικούς φορείς με επαρκείς πόρους και δυναμικό. Στην τροπολογία 586 ε, λέω ότι το προσωπικό θα πρέπει να συνδέεται με τις ανάγκες της αγοράς και να ποικίλουν ανάλογα με αυτές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Επίσης, οι φορείς αυτοί θα πρέπει να αναλαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με προσφυγές ή και κατόπιν δική της ε, πρωτοβουλίας ε, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές που πρέπει να επιληθούν στην αγορά. Επίσης, ε, οι ε, εθνικές αρχές θα πρέπει να ε, τηρούν μητρό των αποφάσεων του, το οποίο να είναι προσβάσιμο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, σημαντική είναι η τροπολογία 591 που έχει να κάνει με τη διαδικασία διορισμού. Η κυρία Μπιλμπάου και εγώ προερχόμαστε από περιφέρειες με ισχυρά κοινοβούλια, με νομοθετικές ε, και δημοσιονομικές ε, αρμοδιότητες και γι' αυτό αλλάξαμε την λέξη Εθνικό Κοινοβούλιο σε αρμόδιο κοινοβούλιο στο άρθρο αυτό όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων από τους ρυθμιστικούς φορείς και την ε, τροπολογία 601 ε, προτείνω δύο εβδομάδες για τη λήψη αποφάσεων. Ε, πιο χρήσιμη όμως είναι η πρόταση του κυρίου Κράμερ για τις 20 εργάσιμες ημέρες. Θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί του. Η τροπολογία 421 προτείνει οι ρυθμιστικές αρχές ε, θα πρέπει να προτείνουν εναλλακτικέ λύσει μαζί με όλου του ενδιαφερόμενου. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό για μα. Ε, και επίση ε, προτείνω στην τροπολογία 619 ο ρυθμιστικό φορέα δύο φορέ το χρόνο να συμβουλεύεται με του προσώπους των χρηστών των σιδηροδρόμων ώστε να λαμβάνει υπόψη του τι δικέ του απόψει. Όσον αφορά την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στην ε, τροπολογία 617 ε, προτείνω τη δυνατότητα προσφυγής προς την Κομισιόν σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών και αυτό είναι σημαντικό για μας. Και επίσης στην τροπολογία 625 προτείνω οι, εθνικές, οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την εργασία τους, την λήψη αποφάσεων και τις πρακτικές που χρησιμοποιούν. Και επίσης η, η Κομισιόν θα πρέπει να διασφαλίζει την ε, αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων. Όσον αφορά ε, τον, ε, έναν Ευρωπαίο ρυθμιστή, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση σύντομα. Ξέρω ότι κάποιοι συνάδελφοι, ο κύριος Γκρός και άλλοι προτείνουν πέντε χρόνια. Ωστόσο μιλάμε για αναδιατύπωση εδώ πέρα, γι' αυτό οι ρυθμιστικοί φορείς ε, θα πρέπει να ε, αρχίσουν να λειτουργούν, οπότε δεν μπορούμε να χάσουμε τόσο χρόνο. Όσον αφορά τη συζήτηση για το unbundling, ε, την αποσύνδεση, συμφωνώ με την ιδέα ότι η... Θα πρέπει να διασφαλίζεται ο, ο διαχωρισμός των λογαριασμών και επίσης ε, δεν, ε, ε, κάποιοι δημόσιοι πόροι που έχουν δοθεί για έναν τομέα δραστηριοτήτων δεν θα πρέπει να μεταφέρονται σε άλλον. Όσον αφορά τις τροπολογίες 654 και 655, έχω ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να επιμείνω, όπως είπε ο κύριος Σοκούν. Δεν θέλω να καταστρέψω τα συστήματα που λειτουργούν καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θα συμφωνήσω με την πρόταση να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει την αγορά και να εξετάσει τις δομές, να εξετάσει τα υπέρ και τα κατά ε, και των δύο διαφορετικών μοντέλων που υπάρχουν. Χωρίς τέτοια ε, επιστημονικά και εμπειρικά στοιχεία θα είναι δύσκολο για μένα να στηρίξω όλες τις τροπολογίες που ζητούν απόλυτο διαχωρισμό ανάμεσα ε, στην διαχείριση των των, ε, ε, των υποδομών ε, και των λειτουργών. Επίσης, τέλος, όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της ανδιατύπωσης, στην τροπολογία 646 προτείνω τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τον νόμο μέχρι Εντό 12 ε, μηνών από την θέση σε ισχύ αυτής της οδηγίας. Ε, το Συμβούλιο ζήτησε 18 μήνες, ε, Χώρε όπως η Ισπανία ζήτησαν 5 χρόνια, για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Και τελευταία παρατήρηση, και εγώ είμαι υπέρ των πινάκων αντιστοιχίας και ελπίζω ότι δεν θα αφαιρεθούν από την αναδιατύπωση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ζήλα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Σεζίλε, θα ήθελα να... Θα ήθελα να ευχηθώ ότι καλύτερο στον ε, εισηγητή μας. Είναι δύσκολο το θέμα, είμαστε ε, ε, βέβαιοι όμως ότι θα προοδεύσει το θέμα αυτό. Ε, η ιδέα του Συμβουλίου ουσιαστικά αποτελεί οπισθοδρόμηση σε σχέση με τα όσα έχουμε συμφωνήσει μέχρι στιγμή. Εμεί θα θέλαμε ε, μια πιο φιλόδοξη λύση. Τώρα θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και να βρούμε καλό συμβιβασμό εντός της Επιτροπής μας και τελικά στην Ολομέλεια. Και γι' αυτό ίσως αυτά που λέω τώρα να διαφέρουν κάπως από αυτά που θα έλεγα εάν δεν υπήρχε, αν δεν γινόταν τελικά αναβολή της ε, συζήτησης. Οι εθνική Νομοθέτη και φορεί θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε και ε, είμαι υπέρ της ιδέας αυτής ε, και σίγουρα και πιθανότατα θα αποτελέσει μέρος συμβιβασμού όσον αφορά τις ε, υπηρεσίες και τις δυνατότητες ε, για τις ε, σιδηροδρομικές εταιρείες, θα πρέπει να πω ότι σε περιπτώσεις όπου προβλέπεται η αποσύνδεση, το unbundling, θα πρέπει να σας θυμίσω το παράδειγμα από τον τομέα των αερομεταφορών στην Γερμανία. Οι υπηρεσίες εδάφους της Lufthansa εξυπηρετούν και άλλες επιχειρήσεις, όχι μόνο την Lufthansa. Θα μπορούσαμε λοιπόν να εφαρμόσουμε αυτήν τη λύση και στους σιδηροδρόμους. Όσον αφορά ε, ένα άλλο θέμα το οποίο μπορεί να μην είναι τόσο επίκαιρο για άλλες χώρες, σίγουρα όμως είναι για τις ε, χώρες της Βαλτικής, ε, όλες οι λύσεις που σχετίζονται με τα σημεία 31 και 32 όσον αφορά την πρόσβαση δηλαδή στις υποδομές και τα όρια. Θα ήθελα να βρούμε καλό συμβιβασμό ανάμεσα στην πρόταση τη δική μου και του κυρίου Μπαλτσίτης. διότι ε, στις χώρες μας έχουμε πολύ καλή αναλογία επιβατών και ε, εμπορικών φορτίων και αυτό είναι Τα εμπορικά φορτία είναι σημαντικά για μας. Θα ήθελα λοιπόν ε, να υπάρχουν εδώ δύο κριτήρια. Από τη μία θα πρέπει να καλύπτεται το κόστος Θα πρέπει να διαμορφώνεται δηλαδή η τιμή της αγοράς, δεν θα πρέπει όμως ε, να είναι χαμηλότερη από το κόστος. Άλλο σημαντικό θέμα ε, είναι η ασφάλιση των φορτίων. Υπάρχουν κάποιες μικρές επιχειρήσεις οι οποίες ε, είχαν στο παρελθόν μονοπόλιο που μπορούν να προσφέρουν ε, υπηρεσίες. υπηρεσίε. έχουμε τις σχετικές τροπολογίες 112 και 484. Έχω και κάποιες ε, όσον αφορά τη στρατηγική. Νομίζω ότι καλό θα είναι να ε, επιτύχουμε συμβιβασμό για παράδειγμα για τα θέματα τα οποία δεν είναι σημεία κλειδιά. Νομίζω χρήσιμο λοιπόν θα ήταν να πετύχουμε συμβιβασμό πρώτα στα επιμέρους θέματα και κατόπιν να φτάσουμε στα σημαντικά. Η αποσύνδεση σίγουρα θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικά θέματα στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Κύριο Κράμερ, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ για την έκθεση, αλλά από συνεργασία έχω δει και καλύτερα. Μας ε, απέκλεισαν από τη συζήτηση συμβαστικών τροπολογιών που επαστέρισαν στου άλλου αλλά όχι σε εμά. Την επομένη μόνο έλαβα τη σχετική ενημέρωση, δηλαδή δεν εκφράζουν εμά συμβαστικέ τροπολογίε και πρέπει να πω ότι όταν συζητούμε αυτά τα θέματα, λέμε στα σημαντικά σημεία ότι είναι απαραίτητα τα αριθμιστικά σώματα, η διαφάνεια και η πρόσβαση για τον καθέναν πολύ σημαντικά θέματα και εντάξει, συμφωνούμε σε αυτά τρία σημαντικά για την αποδέσμευση διαφοροποιούμαστε. Πολύ καλά. Ερωτώ λοιπόν γιατί επιβάλλεται αυτή η πίεση χρόνου και περί τίνος πρόκειται εν τέλει. Είχαμε καταστήσει σαφέ σε μια επιστολή ότι δεν είναι ανοιχτά τα δίκτυα των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη. Από 1η του 2007 το δίκτυο έχει ανοίξει για τις συνδρομικές μεταφορές τυπικά αλλά δεν ε, ισχύει ουσιαστικά και βλέπουμε ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικές τοποθετήσεις. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι ξαφνικά επιβάλλον, ασκούνται πιέσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κοιμόταν επί 9 χρόνια, ξαφνικά ξύπνησε και μας πιέζει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε αποφάσεις. Γιατί? Προφανώς αυτό σχετίζεται με τη διαδικασία επί την οποία έχετε εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου και φαίνεται ότι φοβάστε πως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν θα ακολουθήσει τις, τα δικά σας επιχειρήματα και φοβάστε μήπως και εμείς ε, και θεωρείτε ότι πρέπει πια να αναλάβετε δράση. Ε, αυτό είναι μάλλον ο λόγος αυτών των πιέσεων που μας ασκούνται. Αλλά δεν είναι δική μας δουλειά, σας βγάλουμε από τη δύσκολη θέση. Το δικαστήριο αποφασίζει με βάση την νομοθεσία του 2001. Είτε πρόκειται για, για, για γερμανικό, για γαλλικό ή για ισπανικό μοντέλο, πρέπει να είναι σύμφωνο με τα κείμενα τα νομοθετικά και τις διαδικασίες του 2001. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το αποφασίσω. Δεν μπορώ να το κρίνω γιατί δεν είμαι και νομικός. Γι' αυτό υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μόλι ληφθεί η απόφαση και στη συνέχεια αυτή τη αποφάση θα καταβληθούν οι προσπάθειε έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ε, των σιδηροδρομικών μεταφορών. Θεωρητικά. Αλλά βλέπουμε ξαφνικά δηλώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2006 μάλιστα να επανέρχονται ε, πολύ πιο ριζικές από του 2001 πρέπει να πω προσπαθώντας να διευκρινίσουν τις ρυθμίσεις του 2004, γιατί φαίνεται ότι εκεί πέρα έχουν γίνει τα σφάλματα και υπάρχει κίνδυνος να μας, ε, καταδικάσει, να σας καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ερώτω λοιπόν, εάν αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί δεν, το, δεν με ρημνήσατε να ρυθμίσετε τα ζητήματα αυτά μέσα στην έκθεση, αφού εσείς είστε το μόνο όργανο που έχει το, την εξουσία της πρωτοβουλίας, το δικαίωμα της πρωτοβουλίας, το κοινοβούλιο, του Συμβούλου έχουν δικαίωμα το πρωτο... της Εγώ δεν βλέπω τίποτα για την αποδέσμευση μέσα στο κείμενο της Επιτροπής. Αλλά προφανώς υπάρχει μία λύση ε, διαφοροποιημένη, μία τοποθέτηση διαφοροποιημένη σε επίπεδο επιτροπή. Άλλοι λένε ναι στο unbundling και άλλοι όχι. Γι' αυτό δεν τα έχετε καταφέρει να τα διατυπώσετε σε, με ενιαία γραμμή μέσα στο κείμενο του Κοινοβουλίου. Και υπάρχουν κάποιοι από το Κοινοβούλιο που παίζουν το παιχνίδι αυτό και που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τι δικέ σα επιδιώξει και μέσα από την έκθεση αυτή να επηρεάσουν ε, και να ακολουθήσουν ε, ή να, προλάβουν μάλλον τις εξελίξεις επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όχι. Το θέμα είναι οι συζητήσει οι οποίε έχουμε πραγματοποιήσει είναι, ήταν απόλυτα ξεκάθαρε ότι ανεξάρτητο του αν θα αποφασιστεί η αποδέσμευση ή όχι, δεν θα επηρεαστούν τα ε, δίκτυα και το άνοιγμα των δικτύων. Αλλού μπορεί να υπάρχει πιο έντονη ε, διαδικασία του unbundling και αλλού όχι. Εν γέννη στην Ισπανία Φερρυπίν ισχύει το σύστημα του close shop. Μόνο ένα τρένο νομίζω πάει από την ε, Ισπανία κατευθείαν, περνάει τα σύνορα και πάει στη Γαλλία. Εν γέννη ισχύει το close shop. Αλλού είναι διαφορετικέ συνθήκε. Και έχουμε πει ότι αν συμφωνήσουμε σε αυτά, ανοίγουμε, ανοίγουν τα δίκτυα αμέσω και, και ισχύουν για όλου οι ίδιε συνθήκε πρόσβαση στα δίκτυα. Αλλά φαίνεται ότι κάτι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Εδώ ακριβώ λοιπόν είναι το καθοριστικό σημείο. Πρέπει να λάβουμε γρήγορα αποφάσει και εδώ ακριβώ. Επί της αρχής εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην απόφαση στη Γερμανία, πρέπει να ληφθεί απόφαση μέσα 14 μέρες. Στην Ιταλία μέσα δύο μήνες, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που δεν πληρούνται, άρα θα χρειαστούν και δύο χρόνια ακόμη θα έχει εντωμεταξύ καταστραφεί οικονομικά ο νέο επιχειρηματία που θέλει να μπει στο δίκτυο κτλ. Στη Γαλλία άλλε συνθήκε. Αυτό λοιπόν ε, δείχνει ότι χρειάζεται να έχουμε ρυθμιστική αρχή, ισχυρή ρυθμιστική αρχή στέναρη, η οποία αποτελεί στη τελευταία ανάλυση την θετικότητα των εκφανών για να λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Και στη διαφάνεια που ανέφερε και ο κύριο Κούν, και δεν καταλαβαίνω γιατί το λέτε αυτό, γιατί θα πρέπει να αποσύρετε κάποια τροπολογία η οποία είναι ακριβώ αντίθετη με αυτά τα λόγια που ακούσαμε από το στόμα σα σήμερα στη συνεδρίαση. Διαφάνεια λοιπόν και παροχή τη υπηρεσία που είναι καθοριστική σημασία ιδιαίτερα για το η νέα επιχείρηση που μπαίνει στην αγορά και έχει να ανταγωνιστεί τι παλαιότερε και πρώην κρατικέ επιχειρήσει. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να αποδυναμωθεί ο η ρυθμιστική αρχή. Αυτό δεν το έχουμε πει εμείς. Έχουμε πει αντιθέτω ότι εάν ε, θέλει να χρησιμοποιήσει Φερρυπίν κάποιες εγκαταστάσεις ο νέος στην αγορά. Και το απαντάνε, Α, κοίταξε, δεν υπάρχει χώρος για σένα. Τότε θα πρέπει η ρυθμιστική αρχή να είναι σε θέση να παρέμβει ακόμη και εκεί για να του βρει χώρο, εγκαταστάσεις, θέσεις κτλ. Αυτό πρέπει να επισημάνουμε και νομίζω ότι αν έχουμε αυτά τα τρία σημεία μπορούμε να καταλήξουμε σε καλή συμβαστική απόφαση, τροπολογία, ασκώντας έτσι πίεση προς την κατεύθυνση αυτή. Και αυτό ανεξάρτητα με το unbundling. Όλα τα άλλα τα έχετε ξεκινήσει εσείς. Ευχαριστώ κύριε Βίλς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερα σημεία που είναι σημαντικά για μένα. Καταρχάς, για την τροπολογία 206 για τις υπηρεσίες, όπου νομίζω ότι η ε, διαγραφή της τροπολογίας 22 έχει μεγάλη σημασία. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με την πρόταση για ε, διαρκή και βιώσιμη αποδοτική λειτουργία των μεταφορών που δεν θα πρέπει να αποκοπούν από την αποτελεσματική, από την ουσιαστική λειτουργία των σιδηροδρόμων. Στην, ε, στις επισκευές ε, οι ενοποιημένες ε, επιχειρήσεις συνδρομικών μεταφορών θα μπορούσαν προς το συμφέρον του πολίτη του επιβάτη να βεωσούν εφόσον οργανωθούν αποτελεσματικά ουσιαστικές λύσεις για, το σιδηρόδρομο η διατήρηση και η ανάπτυξη της σιδηροδρομικής επιχείρησης έχει πολύ μεγάλη σημασία όπως αναφέρει και ο σχετικός σύνδεσμος των συνδικάτων των σιδηροδρομικών ε, και έτσι ο διαχωρισμός ε, των υποδομών και της λειτουργίας μπορεί να έχει απρόβλεπτε συνέπειε για τη λειτουργία των γερμανικών σιδηροδρόμων, για την ε, επιβίωση του ομίλου του ίδιου, αλλά και για την διαφύλαξη μια ορθολογική δομή στι μεταφορέ μα. Και βέβαια σε σχέση και με τι ε, περιβαλλοντικέ μα ανησυχίε, τη χρήση των ορεικτών καυσίμων και, άλλες, ε, και επιβολή λύσεων άλλων από το σιδηροδρόμο που είναι ο πιο οικολογικό, ω γνωστόν. Ανησυχίε λοιπόν σχετικέ με την επιβίωση του ομίλου των σιδηροδρόμων τη Γερμανία. Ε, που δείχνουν ότι η γερμανική κυβέρνηση ε, θα πρέπει να κάνει επιλογές ε, ουσιαστικές και μεγάλες τομές. Επίσης, η διαφύλαξη της ελάχιστης υπηρεσίας όπως προτείνουν ορισμένες τροπολογίες εδώ ε, και ο περιορισμός ως εκ τούτου του δικαιώματος στην απεργία είναι για μας απαράδεκτος. Το δικαίωμα της απεργίας είναι ένα ουσιώδες δικαίωμα. Ο χάρτης των ανθρωπινών δικαιωμάτων, όπως λέει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το προβλέπει στο άρθρο 11 και ε, ορίζει ότι μπορεί μόνο για πολύ συγκεκριμένους λόγους να περιοριστεί το δικαίωμα στην απεργία που είναι όπως είπα θεμελιώδες για πολλά από τα στάγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το ε, περιστείλει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει σχετικές αρμοδιότητες περιστολής, άρα μόνο το εθνικό δίκαιο μπορεί να επιβάλλει τέτοιους περιορισμούς. Όπως προβλέπετε στο Αυστριακό Φερρυπίν Εθνικό Δίκαιο υπάρχουν και άλλα έγγραφα διεθνούς ε, χαρακτήρα που προβλέπουν αντίστοιχε ρυθμίσει. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διαγραφεί και να μην αντικατασταθεί από άλλη σχετική τροπολογία περιορίσει το δικαίωμα στην απεργία. Επίση, Θέλω να, να αναφερθώ στις ε, ε νομοθετικές πράξεις, στην οτιολογική σκέψη 65, απορρίπτουμε τις ε, ε, προτάσεις, διότι αυτές ακριβώς είναι εκείνες οι οποίες πλήττουν την ίδια την ουσία της ε, ε λειτουργίας των σιδηροδρόμων και μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρά προβλήματα νομικά, πολιτικά, αλλά και δημοκρατικά, δημοκρατικές λειτουργίες, ο δημοκρατικός έλεγχος και η διαφύλαξη των δημοσίων αγαθών, η στάθμιση δε αυτών ε, θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο αντικειμονικό και όχι ε, συμφεροντολογικό με συμμετοχή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην όλη διαδικασία για την παραγωγή των σχετικών νομοθετημάτων. Και θα ήθελα να ε, σημειώσω για την κυρία Σαρακιάνη και τις λοιπές τροπολογίες τις σχετικές ε, με την ε, επεξεργασία των λεγόμενων συμβαστικών τροπολογιών. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να φτάσουμε στο τέλος της ενοποιημένης και τεχνικά προηγμένης συνδρομικής δικτύωσης, συνδρομικών δικτύων βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο σαν προοπτική και γι' αυτό απορρίπτουμε κάθε σχετική τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν και θα ήθελα να πω ότι ε, υπάρχουν και άλλοι ευρωπαϊκοί σιδηροδρόμοι εκτός από την Deutsche Bahn, τους γερμανικούς σιδηροδρόμους. Προχωράμε τώρα στους άλλους ευρωβουλευτές ο κύριος Γκρός, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Και θα ήθελα να της ευχηθώ και κουράγιο για το μέλλον. Ελπίζω να μην ε, θέλει να υποβάλει ο καθένα εδώ πέρα τις ε, απόψει που αφορούν ε, του σιδηροδρόμου τη χώρα του. 27 κράτη-μέλη έχουμε. Ελπίζω ότι θα μπορούμε να σκεφτούμε ευρωπαϊκά, γνωρίζοντα ότι ό,τι έχουμε στην πατρίδα μας δεν είναι απαραίτητα ό,τι καλύτερο για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ και 10 χρόνια θέλουμε περισσότερους επιβάτες και περισσότερα εμπορικά φορτία στους σιδηροδρόμους, γι' αυτό χρειαζόμαστε καλύτερη υποδομή. Θέλουμε επίσης σωστές τιμές, θέλαμε καλύτερη κατάρτιση, αμοιβαία αναγνώριση της κατάρτισης, που σημαίνει επίσης ότι δεν θέλουμε ε, ε χαμηλές αμοιβέ, θέλουμε καλά εκπαιδευμένους ανθρώπους στον τομέα αυτό. Και τώρα ε, θέτουμε το ερώτημα πώς το έχουμε πετύχει αυτό. Και ε, αυτό είναι ε, για μένα το βασικό ερώτημα που πρέπει να θέσουμε. Δεν έχουμε πετύχει τους στόχους αυτούς, ε, σίγουρα όχι. Και δεν τους έχουμε πετύχει, διότι αυτά τα οποία είπαμε δεν έγιναν σεβαστά σε καμία χώρα. Και τώρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα Φτάνουν κάποια κράτη-μέλη ε, στο συμπέρασμα ότι ε, θα έχουμε λιγότερους ανθρώπους ε, και φορτία στους σιδηροδρόμους και ότι θα έχουμε και πολύ χαμηλές αμοιβέ. Αυτό γίνεται όμως ακριβώς χωρίς το ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς θέλουμε να είναι αποτελεσματικοί σιδηροδρόμοι, θέλουμε να υπάρξουν επενδύσεις και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Όποιος σκέφτεται μόνο εθνικά θέλει ακριβώς το αντίθετο. Ε, και αυτό είναι και υπονοούμενο σχετικά με το τι συμβαίνει στο Συμβούλιο. Ε, οι υπουργοί μα δεν δίνουν ελπίδα στου σιδηροδρόμους, δεν δίνουν την ευκαιρία στου σιδηροδρόμους να αναπτυχθούν. Εάν του δίνανε μια ευκαιρία δεν θα είχαμε πια αυτούς τους 6.000 ε, κανόνε, διότι σε, ευρω... σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να αναθέσουν σε μια υπηρεσία τα θέματα αυτά και έτσι δεν ε, θα είχαμε αυτή τη δυσκολία στην αμοιβαία αναγνώριση. Και τι μπορούμε να κάνουμε στους άλλους τομείς. Σίγουρα μπορούμε να φροντίσουμε ε, η διαχείριση των υποδομών ε, αύριο όχι μόνο να, γίνει, να χρηματοδοτηθεί σωστά, αλλά να είναι και οι συνθήκες όμοιε για όλου. Αυτό απαιτεί διαφάνεια όμως και όποιο θέλει διαφάνεια ε, δεν θα πρέπει να ανησυχεί κιόλα για τον έλεγχο και για, ακριβώς γι' αυτό χρειαζόμαστε έναν ε, ισχυρό ε, ρυθμιστή, όχι... Ελπίζω να μην καταλήξουμε σε καταστάσεις όπως βλέπουμε στο ποδόσφαιρο. Τέλος, θα ήθελα επίσης να πω, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, ότι δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς ε, εάν έχει ε, ε, δημόσιο χρήμα. Καλά, συγγνώμη, στην Ιταλία είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ε, όποιος, λέω, όταν μιλάμε για τις υπηρεσίες, δεν θα πρέπει να ανησυχούμε όταν απαιτείται διαφάνεια τη στιγμή που ε, χρησιμοποιούνται δημόσια χρήματα και δεύτερον, όταν είναι δικαιολογημένο το ερώτημα. Ε, τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για να βελτιωθεί η ε, υποδομή ή για να ε, βοηθήσουν τους, τους οικονομικούς φορείς για να είναι πιο ανταγωνιστικοί. Εάν λοιπόν έχουμε σωστή απάντηση στα ερωτήματα αυτά, αυτό θα ωφελήσει τους σιδηροδρόμους και θα βρούμε ένα θα καταλήξουμε σε μία λύση όπου η αποσύνδεση θα ε, είναι δικαιολογημένη, διότι σήμερα, και θα μπορούσα να ε, σας προβάλλω και άλλα επιχειρήματα, είμαι πεπισμένος ότι καμία χώρα δεν μπορεί σήμερα να δικαιολογήσει, η υπηρεσία ε, λειτουργίας να επηρεάζει την ε, υποδομή και να αποφασίζει και ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί την υποδομή αυτή. Θα πρέπει να υπάρξει αποσύνδεση, αλλά θα πρέπει σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο να ε, παράσχουμε όλες αυτές τις εγγυήσεις και όχι αντίστροφα. Ευχαριστώ. Uh, Ο κύριος Αλκαντράου, αν μπορείτε να περιοριστείτε στα τέσσερα λεπτά θα είμαι ευγνώμων. Θα κάνω ό,τι μπορώ κύριε Πρόεδρε. Ε, τεχνικά είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα αυτό και πολιτικά είναι δύσκολο. Ε, εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία για τους επόμενους μήνες. Θα πρέπει εδώ να καταστήσουμε σαφές ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε κάτι το οποίο να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε, ώστε ε, οι ευρωπαϊκοί σιδηρότρομοι να γίνουν αποδοτικότεροι και ε, κάτι που θα ωφελήσει τους καταναλωτές ε, και τους εργαζόμενους στον τομέα. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για το ρυθμιστικό φορέα, όταν μιλάμε για το δυναμικό, θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα ακόμα πιο πέρα. Ε, κάποια προβλήματα όπως οι επιπτώσεις στην αγορά θα πρέπει να έχουν την ίδια ερμηνεία στα διάφορα κράτη-μέλη και θα πρέπει να εξετάσουμε μήπως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα προστάδιο του Ευρωπαϊκού Ρυθμιστικού Φορέα, για παράδειγμα για τις ε, μεταφορές εμπορευμάτων. Επίσης, πώς μπορούμε ε, καλύτερα να διασφαλίσουμε τους ε, πόρους για την υποδομή. Θα χρειαστούμε δισεκατομμύρια. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι να ακολουθήσουμε την εισηγήτρια. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες πτυχές. ποιες δαπάνε μπορούν να αντισταθμιστούν και πώς. Και ένα ακόμα θέμα. Ίσως θα πρέπει να το εξηγήσω αυτό. Οι τιμές ποικίλουν πολύ στα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω αν αυτό ε, είναι δικαιολογημένο. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια για, την, για τον υπολογισμό των τιμών. Και όσον αφορά την αποσύνδεση, η συγκήτρια έχει προσπαθήσει να βρει ε, συμβιβασμό ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν ε, απόλυτη αποσύνδεση, unbundling, και αυτούς που δεν το θέλουν. Θα πρέπει ίσως να συζητήσουμε πώς... Ε, πόσο οξία είναι η διατύπωση, μήπως ε, πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα των ε, σημαντικών υπηρεσιών. Όλοι θέλουμε ο διαχειριστής των υποδομών να είναι ανεξάρτητος και όλοι οι οικονομικοί φορείς να έχουν την ίδια πρόσβαση στην υποδομή. Και όσον αφορά τις μεταφορές επιβατών, πριν ένα χρόνο, όταν ψηφίσαμε το τρίτο σιδηροδρομικό πακέτο, συμφωνήσαμε και με τα άλλα θεσμικά όργανα να έχουμε τη συζήτηση αυτή το 2012 και ε, ε, η Κομισιόν ε, θα υποβάλει σχετική πρόταση. Δεν θα πρέπει να προδικάσουμε τα αποτελέσματα, θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ντουιρόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την περίληψη που μας παρουσίασε, που όμως αποτελεί περίληψη των διαφόρων τροπολογιών. Εγώ δεν είδα, δεν διαβλέπω μια γραμμή, μια τοποθέτηση που θέλει να περάσει μέσα από την έκθεσή της η εισηγήτρια. Και είναι λυπηρό αυτό, γιατί καθήκον δικών μας είναι της Επιτροπής μας των Κοινοβουλευτών πολιτικών εκπροσώπων που είμαστε εμεί, να διατυπώσουμε μια γραμμή γιατί βέβαια ξέρουμε ότι το Συμβούλιο δεν πρόκειται να ε, βοηθήσει στην σύσταση ενό ευρωπαϊκού συνδρομικού χώρου γιατί κάθε χώρο θα δραβεί προ τη δική τη κατεύθυνση. Θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα σημεία που ξεκινούν από αυτά που είπε και ο κύριο Κράμερ εμβάθυνση υποδομές, διαχωρισμός είναι βέβαια βασικές αρχές ε, στις οποίες δεν χρειάζεται να τοποθετηθώ περισσότερο. Δεν χρειάζεται να εμβαθύνουμε δηλαδή την, ε, ε, το διαχωρισμό εκτός βέβαια από τον οργανωτικό, από, τις, από την παροχή των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Ναι, στην περισσότερη διαφάνεια και τη σχέση μεταξύ των διαφόρων συνιστοσών του συστήματος, οργάνωση σε εθνικό επίπεδο, γιατί εκεί νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό καλύτερα και στις περιπτώσεις η ρύθμιση γίνεται σε εθνικό επίπεδο, αλλά με τη δυνατότητα της διαιτησίας της Ευρωπαϊκής, αν προκύψει πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κλωτσίσουμε τη φωλιά των τερμητών και να ελπίζουμε στη συνέχεια ότι αφού ξεσπάσει το κακό θα ξαναπέσουν τα κομμάτια ένα-ένα στη θέση του και θα ανασυσταθεί το μοσαϊκό εάν αποφασίσουμε να ανατρέψουμε τους χρόνους του παιχνιδιού, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Επίσης λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να δεχθούμε ότι δεν είναι δυνατόν οι ιστορικοί ε, φορείς ε, και χειριστές να εκδιωχθούν ανεφετέρου ε, από τα συστήματα που διαχειρίζονται. Πρέπει να έχουμε και λογική και πρόνοια στην υπόθεση αυτή και προνοητική στάση. Αυτός ε, ο φάκελος δεν έχει να κάνει μόνο με τεχνική αναδιαμόρφωση, αποτελεί ένα ζήτημα πολιτικής και μηνυμάτων που θέλουμε να αποστείλουμε και για την οργάνωση, νέα οργάνωση με σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων, αλλά όσο δυνατόν πιο αποτελεσματική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που να μην είμαστε κολλημένοι ο καθένα στην ιδεολογία του, αλλά να προχωρήσουμε μέσα από συστήματα τα οποία να μα φέρουν προ το μέλλον Ξέρω ότι η συγγήτρια έχει πολλά θέματα να διαχειριστεί και πολλές τροπολογίες, αλλά σημαντικό θα ήταν να έχουμε ένα μήτο της για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε που βαίνει αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και δεδομένου ότι το Συμβούλιο ξέρουμε ότι είναι προσκαλυμμένο στα εθνικά συστήματα, ενώ από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπόρεσε να κρίνει και να λάβει τις στεναρές θέσεις που όφιλε. Άρα θα πρέπει να το πράξουμε εμεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο μια ευθυγράμμιση των τροπολογιών σε τεχνικέ προσαρμογέ που στη τελευταία δεν προσφέρουν και τίποτα. Ο Πρόεδρο. Θα ήθελα να σημειώσω ότι υπάρχουν αρκετέ συμβαστικέ τροπολογίε εδώ μεταξύ. Να σου πω, Μάικλ, κοίταξε, να επικοινωνήσει με το, να δεις ε, τι σύστημα επικοινωνία έχει η ομάδα σου, πως εκεί είναι το πρόβλημα και γι' αυτό δεν ενημερώνεσαι. Όχι, υπάρχουν συμβαστικέ τροπολογίες και κάποιοι τις επεξεργάζονται. Είναι σκληρό να επιτίθεται κανεί ε, κατά ε, εισηγητή που έχει 750 τροπολογίες να διαχειριστεί και να λένε «Α, δεν με ενημέρωσε και δεν ξέρω» και τέτοια. Είναι λίγο υπερβολικέ σκληρέ αυτέ οι επικρίσει. Φυσικά προ, προσέχουμε ότι δουλειά κάνει η συγγήτρια να γίνεται κατά τρόπο συμπεριληπτικό ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλε οι ομάδε. Κύριο Κάντσιαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει. Να πω ότι είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό, είναι πολιτικά φορτισμένο. Έχουμε κάποιο χρόνο ακόμα, έχουμε όμως και πάρα πολλή δουλειά μέχρι τότε. Πολύ συχνά παρουσιάζουμε τις θέσεις μας ε, και λέμε ότι το Συμβούλιο δεν τα θέλει αυτά. Είναι σαν να λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση αυτά που θέλει το Συμβούλιο. Εγώ νομίζω όμως ότι θα πρέπει να ε, πετύχουμε περισσότερη συνένεση ε, εδώ εντός του Κοινοβουλίου. Έχω εδώ κάποιες προτάσεις για να έχουμε καλύτερη απελευθέρωση, αποσύνδεση και όσον αφορά τον ρυθμιστικό φορέα. Καταρχήν, ε, όσον αφορά την ε, απελευθέρωση της αγοράς, εάν δεν απελευθερωθεί η αγορά ε, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο στόχος, γιατί δυσκολεύουμε τη ζωή μας εάν δεν έχουμε στόχο να επιτρέψουμε στον κόσμο να ταξιδεύει σε, στα πλαίσια ενός ενιαίου σιδηροδρομικού συστήματος. Επίσης, έχουμε κάποιες οδηγίες σχετικά με τις ε, δημόσιες κοινοφιλείς υπηρεσίες. Ε, ε, ίσως θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε κάποιες... Ίσως μπορούσαμε να επιβάλλουμε κάποιους κανόνες στο περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αυτός θα πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος μας. Και όσον αφορά το τέταρτο πρόγραμμα δεν ε, είμαι βέβαιος γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε ήδη αυτό το επόμενο στάδιο. Εάν 12 μήνες ε, δεν ε, αρκούν, τότε ίσως θα μπορούσαμε να παρατείνουμε το χρονικό διάστημα και στόχος είναι να έχουμε σε όλα τα κράτη-μέλη ιδίου τύπου υπηρεσίες. Να έχουμε μία συμβαστική ανάμεσα στις ε, σωστές κατευθύνσεις ώστε να μπορέσουμε εκτός από το να, να ελέγξουμε τους διορισμούς ε, για όσον αφορά το ποιο ασκεί την... τον έλεγχο στις υποδομές να πούμε και ποιος ορίζει, ποιος ορίζει αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Έπειτα. Όσον αφορά το ρυθμιστικό φορέα, θα πρέπει θεωρητικά να είναι ευρωπαϊκός, αλλά μεταξύ θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχύσουμε τους ε, εθνικούς μας συντονιστές και να προσπαθήσουμε να τους συνδέσουμε με τον Ευρωπαίο. Τώρα, το κομμάτι που αφορά τις υποδομές, πέρα από τις ε, ράγες, πέρα από όλες τις υποδομές που θεωρούμε απαραίτητε κατά τη διάρκεια των αξένων, θα πρέπει να βελτιωθούν και οι σταθμοί. Οι σταθμοί και όσοι ασχολούνται με τις υποδομές, εν πάση περιπτώσει με εκείνες τις υποδομές που είναι χρήσιμες για να μπορούν να, να περνούν τα τρένα, να περάσουν στο παράρτημα 1 που σχετίζεται με την ιδιοκτησία των υποδομών. Πιστεύω πως η αρχή λοιπόν ήταν λίγο επικίνδυνη, αλλά Τώρα δεν θα πρέπει να υποχωρήσεις, να προχωρήσεις σε αυτά τα σημαντικά θέματα που αφορούν αυτό που είναι η βασική λειτουργία αυτού του φοντοσχέδιου, δηλαδή απελευθέρωση των εθνικών και περιφερειακών ε, επιβατών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Ερτούγκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ομολογήσω ότι όντω δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν είναι και δίκαιο να επικρίνει κανεί ε, την εισηγήτρια σαν να μην ήταν ε, συνεργατική και πρόθυμη να συνεργαστεί. Έχουμε ένα σοβαρό, ένα περίπλοκο σημαντικό, αλλά και συναισθηματικά φορτισμένο θέμα και προσπαθεί να συνδυάσει το δυνατόν περισσότερο τις απόψεις, τις διαφορετικές απόψεις για τη ρυθμιστική αρχή. Για τις ρυθμιστικές αρχές είμαι πεπισμένος ότι έχει κάνει σωστέ επιλογέ η συγκήτρια. Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητε, να έχουν ευρείε αρμοδιότητε και την κατάλληλη. Ε, ε τις κατάλληλες εξουσίες. για τα residential facilities νομίζω ότι θα πρέπει, εφόσον δεν αξιοποιούνται, να μην εκτίθενται σε ε, leasing, προνομίστωση, αλλά σε πώληση. Επίσης, η ελεύθερη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις αγορές θα πρέπει να, είναι, να ισχύει για τους πάντες, σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις συνδρομικές επιχειρήσεις. και το όργανο που θα λαμβάνει τι αποφάσει, διοικητικό συμβούλιο κτλ. θα πρέπει να έχει τι σχετικέ εξουσίε. Αυτό θα πρέπει να μα απασχολήσει τι επόμενε εβδομάδε. Θα πρέπει να βρούμε μία λύση χωρί να ε, κατακριουργήσουμε το ισχύον σύστημα, αλλά να βρούμε μία λογική λύση για να μπορούν να λειτουργούν ουσιαστικά οι ρυθμιστικέ αρχέ. Επίση, οι ε, δομές θα πρέπει να διατηρούνται στο βαθμό που δεν ε, βαίνουν κατά του ελεύθερου ανταγωνισμού. και που δεν ε, είναι αντίθετε με τι βασικέ αρχέ τη ελεύθερη οικονομία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν χώρε οι οποίε έχουν όχι μόνο μη στην επιχείρηση, αλλά πολλέ και μάλιστα οργανωμένε σε σύστημα holding κτλ. Επίσης, δεν μπορούμε να λησμονούμε ότι υπάρχουν συλλογικέ συμβάσει, τουλάχιστον αυτό ισχύει στη Γερμανία και φανταζόμαι ότι και σε άλλε χώρε θα υπάρχει κάτι αντίστοιχο, οι οποίε ε, ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε περίπτωση όπου μπορεί η ε, απελευθέρωση της αγοράς να οδηγήσει σε επιδείνωση των συνθήκων και για την επιχείρηση. Το δικαίωμα στην απεργία, για να ολοκληρώνω, έχει ψηλότερη αξία από τις ελάχιστες ε, παραεχόμενες ε, υπηρεσίες <clears throat> και οι υποδομές ξέρουμε ότι σε όλη την Ευρώπη παρουσιάζουν προβλήματα, άρα θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρότητα και το εάν θα πρέπει να αποκοπούν οι μία από το υπόλοιπο σύστημα. Αλλά όσο δεν είναι οι τιμές προσαρμοσμένες στις ε, συνθήκες, θα έχουμε τίμημα υπερβολικά υψηλό για τον πολίτη, επιβάτη. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα έχουμε το χρόνο μέχρι τον Οκτώβριο να μελετήσουμε πολύ προσεκτικά το θέμα και να καταλήξουμε σε λογικές συμβαστικές τροπολογίες που θα εξασφαλίσουν τον πλουραλισμό και καλή διαχείριση των στερεοδρόμων μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σφιντάντσα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την στήριξή μου στην εισηγήτρια για αυτό πολύ δύσκολο, το πολύ δύσκολο έργο που έχει αναλάβει. Μερικές εβδομάδες παραπάνω Νομίζω θα είναι χρήσιμες για να βρούμε το κατάλληλο πλαίσιο για την συζήτησή μας. Έπειτα, θα ήθελα να τονίσω, όπως και ο συνάδελφος Καντζάν, το θέμα του ανοίγματο των αγορών. Για μένα είναι απόλυτη προτεραιότητα αυτό. Δεν πιστεύω, και το λέω στον συνάδελφο Καντράουι, ότι μπορούμε παθητικά να περιμένουμε το 2012 αναμένοντας πρωτοβουλία της Επιτροπής. Εμείς εδώ ασχολούμαστε με το θέμα της πρόσβασης στις υποδομές. Δεν μπορούμε παρά να δώσουμε μια στεναρή όθηση προς την κατεύθυνση ενός μεγαλύτερου ανοίγματο της αγοράς. Είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να φτάσουμε σε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα, έτσι ώστε να διευρυνθεί η προσφορά και να βελτιωθούν οι υπηρεσίες ε, για τους Ευρωπαίους πολίτε. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να δούμε μέχρι ποια φάση θα το κάνουμε. Ίσως ε, για τι περιφερειακέ ε, μεταφορές να το καθυστερήσουμε ίσως, αλλά για τις εθνικές μεταφορές σίγουρα θα πρέπει να προχωρήσουμε. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο των εθνικών αριθμιστικών φορέων που θα πρέπει να είναι ανεξάρτητε αρχέ με συγκεκριμένε αρμοδιότητε. Γι' αυτό ήδη υπάρχουν θετικέ τροπολογίε και είμαι πεπισμένο ότι η πρόταση τη εισηγήτρια να δημιουργηθεί ένα δίκτυο εθνικών ρυθμιστικών φορέων είναι ένα βήμα μπροστά, με πρόθεση να φτάσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα σε έναν ρυθμιστικό, ευρωπαϊκό μάλλον ρυθμιστικό φορέα που θα υποπτεύεται τους εθνικούς φορείς και θα συμπληρώνει τις ελλείψεις τους, όπως γίνεται και σε άλλους τομείς. Αναμένοντας τώρα την επίτευξη αυτού του μεσοπρόθεσμου στόχου για μια ευρωπαϊκή αρχή, ε, θεωρώ πως μεγαλύτερη συμμετοχή και καλύτερο συντονισμός από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τους εθνικούς ε, ε, ρυθμιστικούς φορείς θα ήταν κάτι το καλό. Τώρα, για την αποδέσμευση, το unbundling, πιστεύω πως ήταν σκόπιμο να συνεχίσουμε σε ένα μερικό ολοκληρωμένο πρότυπο ναι, εξασφάλιση των βασικών ε, υπηρεσιών. Για να εγγυηθούμε την ανεξαρτησία, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξουν χωριστέ αρμοδιότητε, εμπιστευτικότητα των ε, ενημέρωση, μεγαλύτερη διαφάνεια, για παράδειγμα στην διαχείριση του προσωπικού. Όλο ιδιαίτερο είμαι πεπισμένο ότι είναι σημαντικό να επιμένουμε για την ανεξαρτησία, τη διαφάνεια αυτού του τμήματο ε, των ε, διαχειριστών τη υποδομή που ε, διαχειρίζεται την απόδοση των αξώνων και απέναντι στι ομίλου όπου αυτοί υπάρχουν, στα holding. Για να είναι αποτελεσματικό το άνοιγμα της αγοράς θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα την υπόθεση των υποδομών, όπως έλεγε ο συνάδελφος Καντσάν, σε σχέση με το τελευταίο τμήμα και τους σταθμούς που θα πρέπει να επαναταχθούν στην έννοια της υποδομής. Τέλος, οι προτεραιότητες που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι άνοιγμα στην αγορά, ισχυρός ρόλος των εθνικών ρυθμιστικών αρχών μέσα στην προοπτική ενός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα και ε, χωριστές βασικές ε, ε, λειτουργίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Τσικάου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτριά μας για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει και να της ευχηθώ καλή επιτυχία. Τώρα, όσον αφορά τις επενδύσεις στον συνδυοδομικό τομέα, ε, διαπιστώνουμε πως δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το επίπεδο των επενδύσεων έχει πέσει τόσο για τη συντήρηση των υποδομών όσο και για την δημιουργία νέων υποδομών ή τον εξυγχρονισμό της, ε, των υποδομών. Σε ορισμένα κάτι μέλη η ποιότητα των υπηρεσιών έχει πέσει επίσης. Θα θέλ, βλέπουμε όμως ότι αυξάνεται ο αριθμό των επιβατών και ο αριθμό των επιχειρήσεων που μεταφέρουν σιδηροδρομικώς εμπορεύματα. Επίση, το νέο σιδηροδρομικό πακέτο θα πρέπει να αυξήσει την ποιότητα και την ασφάλεια των θέσεων απασχόλησης στον τομέα αυτό. Θα θέλαμε να έχουμε μια αρχή ε, ρύθμισης όσο γίνεται πιο ισχυρή, μεγάλη διαφάνεια, ανταγωνισμό, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Η διάκριση ανάμεσα στη διαχείριση των υποδομών και την εκμετάλλευση των υπηρεσιών μεταφορών θα πρέπει να έχει αρνητικέ επιπτώσει στι συνθήκε απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων στον τομέα. Θα πρέπει να σεβαστούμε τις κοινωνικές ρήτρες ώστε να αποφευχθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ και ο αθέμητος ανταγωνισμός. Και, αν, και εδώ μιλώ κυρίως για νέους φορείς ε, και νέες επιχειρήσεις στην αγορά. Επίση, οι, οι όροι πρόσβαση στι ιδεοδρομικέ υποδομέ δεν πρέπει να έχουν ω συνέπεια την αδυναμία των ε, ταξιδιωτών να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίε που ή να υπάρχει αρνητική επίπτωση στην τιμή των ε, εισιτηρίων. Επιπλέον ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εποπτεύει τις εξελίξεις στον τομέα της απασχόλησης και στις κοινωνικές συνθήκες, καθώς και να σέβεται την, το θεμητό ανταγωνισμό στον τομέα αυτό. Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει σε επαφή με τα συνδικάτα και τις ενώσεις τους, καθώς και τους εκπροσώπους των χρηστών. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του συστήματος των συνδρομικών μεταφορών, θεωρώ πως ήταν σημαντικό. Ακόμα και αν τα κρατημέλη μπορούν να αναθέσουν σε κάποιον συνδρομικό φορέα τη δυνατότητα να συμβάλλει στην ανάπτυξη της των σιδηροδρομικών υποδομών, την ευθύνη να φέρουν πάντοτε τα ίδια τα κρατημέλη. Είναι δηλαδή σημαντικό οι κυβερνήσει να εξασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση και γι' αυτό και πιστεύω ότι σε εθνικό επίπεδο Σε εθνικό επίπεδο, σχεδιασμό ε, για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών θα έπρεπε να είναι δεκαετή. Πιστεύω πως θα πρέπει να δοθεί επίσης απαραίτητος χρόνο στα κράτη-μέλη για να εξυγχρονιστούν και να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο ευρωπαϊκό σύστημα ε, και την προσαρμογή των σειρμών στα ευρωπαϊκά συστήματα. Μιλάω για τις, την 719 και την 720. Έχουμε τα δύο προηγούμενα συντηρητικά πακέτα εντωμεταξύ που δεν έγιναν δεκτά από τα κράτη-μέλη, πράγμα που δεν μας επιτρέπει να έχουμε ε, μια άποψη ανταγωνιστική για αυτή την αγορά. Είναι μια ανταγωνιστική αγορά και είναι απαραίτητο αυτό για να αναπτυχθεί και να αυξηθεί το τμήμα που καλύπτουν οι μεταφορές. Η κυρία Μπιλμπάου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώ να εξηγήσω την γραμμή που ακολούθησε και τις τροπολογίες μου, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να αναπτυχθεί ένας νέος χώρος συνδροδρόμων αποτελεσματικός, λειτουργικός, ε, οικονομικός, διαλειτουργικός, με καλύτερη υπηρεσία για τον επιβάτη, για τον πελάτη εν και γι' αυτό στις τροπολογίες μου ιδιαίτερα ε, με την ιδέα της, του πραγματικού ανοίγματο, της πραγματικής απελευθέρωσης του χώρου των σιδηροδρομικών μεταφορών. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να οργανωθούν ε, με το βέλτιστο δυνατό τρόπο όλες οι φυστάμενες λειτουργίες, πρέπει να γίνει το άνοιγμα μας δυνατόν πιο αντικειμενικές συνθήκες και συνθήκες διαφάνειας, να υπάρξουν επαρκείς ε, επενδύσεις στις υποδομές και να διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα. Επίσης πρέπει να έχουμε ώστε δυνατόν καλύτερο συνδυασμό των επιχειρήσεων, επιχειρήσεων, των υποδομών και την διαφύλαξη των δομών. Η εποπτεία ή εποπτικές αρχές είναι απαραίτητο να έχουν επαρκείς ε, όρους ε, ανεξαρτησίας και εξουσίας για να παρακολουθούν τη λειτουργία του συστήματος. Επενδύσεις χρειάζονται και με μακροπρόθεσμη θεώρηση και σχετικό προϋπολογισμό, με υποστήριξη από όλα τα θεσμικά όργανα και όπως είπε και ο κύριος Τρεμόσα, υποστηρίζω με την τροπολογία 341 την ανάγκη να μεριμνήσουμε ώστε να επιβληθεί η δικασία της διαβούλευσης με τις περιφερειακές αρχές επίδοκρατων κρατών μελών για την για τις εξελίξεις και τις αποφάσεις που θα ληφθούν ε, προκειμένου να ε, γίνουν σεβαστές ε, οι ιδιαιτερότητες στην κάθε περιοχή και περιφέρεια. Άλλωστε οι περιφερειακές αρχές έχουν και ίδιες αρμοδιότητες, έχουν στρατηγικές για τους ιδιαιτεροδρόμους και αυτό το λόγο θα πρέπει να τις εντάξουμε σε αυτές τις προσπάθειες. Και επίσης θα πρέπει να υπάρξει ένας οργανισμός ρυθμιστικός, ευρωπαϊκός, ανεξάρτητος, αποτελεσματικός. Και δυνατόν να θεσπιστεί το χετερό δυνατό, μέσα σε δύο χρόνια και σε πέντε. Μέχρι τώρα θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν βλέπω πουθενά κανένα επιχείρημα ικανοποιητικό γιατί δεν θα πρέπει να ενσωματωθούν ε, οι δομές μέσα στην ε, στο σύστημα εφόσον προσφέρουν ικανοποιητικέ ε, συνθήκες διαφάνειας, ε, αερομικής ασφάλεια. κλπ. Λοιπόν, ο κύριος Ρικέ, ευχαριστώ Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ τη συνάδελφο για τη δουλειά τη. Το μεγάλο δίκτυο είναι, το δίκτυο των σιδηροδρόμων είναι το σύμβολο της Ευρώπης. Συμβολίζει την Ευρώπη και ξέρουμε ότι αυτό ισχύει για τα πάντα στην Ευρώπη, όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές μεταφορές, δηλαδή χρειάζεται και διαφάνεια και ε, ολοκληρωμένα συστήματα και διαφοροποίηση και επενδύσει. Ξέρουμε ότι είναι χρόνια προσπαθούμε, δεν έχουμε φτάσει όμω στο στόχο μα. Όλοι ξέρουμε τι χρειάζεται για να έχουμε ένα αποτελεσματικό, καλά λειτουργούν σύστημα των σιδηροδρόμων. Πρέπει να υπάρξει το άνοιγμα, η απελευθέρωση, η καλή και ισχυρή ρυθμιστική αρχή, ε, η λήψη υπόψη των κοινωνικών συνθήκων, ε, των δημοσίων αγορών. Όλα αυτά είναι στοιχεία και πολιτικά φυσικά, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, αλλά και οικονομικά οι οικονομικέ παράμετροι του συστήματος. Πρέπει να υπάρχουν υποδομές με κατάλληλα μέσα τόσο χρηματοοικονομικά όσο και διαφάνειας. Όλοι γνωρίζουν ποιοι είναι οι όροι. Γιατί λοιπόν να διαφωνούμε δεν καταλαβαίνω. Public holding μου λέτε είναι κάτι που λειτουργεί ικανοποιητικά και δεν χρειάζεται να το ανατρέψουμε. Ναι, αλλά κάθε μονοπωλιακό σύστημα θεωρεί ότι καλά κάνει και υπάρχει και δεν πρέπει να ανατραπεί. Αλλά πρέπει να εξηγήσουμε και γιατί υπάρχουν αυτά τα μονοπωλιακά συστήματα και ποιον εξυπηρετούν. Ε, εάν δεν είναι ικανοποιητική η λειτουργία του, θα πρέπει να τα καταργήσουμε και να τα καταστήσουμε από κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να μένουμε μέσα στα συστήματα αυτά μόνο και μόνο γιατί μα βολεύει να μην αλλάξουμε τίποτα. Και επίση, η εισηγήτρια Ξέρω ότι ασχολείται με θέματα τα οποία δεν ε, βλέπουν διαφοροποίηση μεταξύ πολιτικών ομάδων για λόγους πολιτικούς, αλλά μάλλον για λόγους εθνικούς μεταξύ κάτων μελών. Και ακριβώ εκεί θα είναι το πρόβλημα, ότι αν δεν αλλάξουμε θεώρηση θα μείνουμε στην ίδια κατάσταση που είμαστε ε, και τα τελευταία 15 χρόνια. Και επίσης, σημειώνω ότι όταν είδα τα πρώτα τι ε, πρώτε προτάσει τη Επιτροπής μου είχα αισθανθεί βαθύτερη απογοήτευση. Τώρα βλέποντα τι θέσει του Συμβουλίου ε, οφείλω να ζητήσω συγγνώμη από την Επιτροπή γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πολύ καλύτερε προτάσει από αυτέ του Συμβουλίου και ότι δηλαδή στην πρώτη σιδηροδρόμων ότι να πάμε προ τα μπρο υπάρχει κίνδυνο ακόμη και να πάμε προ τα πίσω. Θα ήθελα επίση να ε, αναφερθώ στην ε, Λευκή Βίβλο, η οποία βλέπει για τα επόμενα 10, 20, 30, 40 χρόνια ε, τις ωραίες μεταφορές, τις ολοκληρωμένες, τις ελεύθερες κτλ. Μας τελευταία να μιλάμε για σιδηροδρόμους κυρίες και κύριοι και εδώ ε, χωρίς να ξέρω φυσικά και να μπορώ να προβλέψω πώς θα καταλήξει αυτό το εγχείρημα στα χέρια του Συμβουλίου, η Λευκή Βίβλο, είπατε κύριε Γκρός, ότι ε, το να μιλάμε σε, για την περίοδο των προσεχών 50 ετών είναι υπερβολικό, αλλά κύριε Γκρόσο, με την κατάσταση που έχουμε δεν είναι νομίζω πολλά τα 50 χρόνια. Ο κύριος Παχ, ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, θα ήθελα να επικροτήσω τις προσπάθειες ε, της συναδέρφου Σαρακιάνη και να της ευχηθώ και κάθε επιτυχία στο μέλλον. Νομίζω ότι οφείλεται στην, ε, στις δικές τους προσπάθειες το ότι έχει καταφέρει να ξεφύγει, να ξεπεράσει την ε, πρόταση της ε, Κομισιόν. Επίσης επικροτώ την αναβολή, διότι έτσι έχουμε περισσότερο χρόνο να αξιολογήσουμε το δύσκολο αυτό θέμα και ότι πιστεύω ότι τους μήνες αυτούς θα πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε ώστε να συζητήσουμε τις συμβαστικές προτάσεις. Πολύ σύντομα να αναφερθώ σε κάποια σημεία με τα οποία δεν συμφωνώ. Ε, έχω υποβάλει και σχετικές ε, τροπολογίες. Ε, όσον αφορά την αποσύνδεση, το unbundling, πιστεύω ότι πρέπει εδώ να συγκεντρώσουμε τις διάφορες εμπειρίες που υπάρχουν, τις διάφορες πρακτικές και επίσης δεν θα πρέπει να έχουμε διακρίσεις και κάτι που με οδηγεί ε, στο, στη δεύτερη μου παρατήρηση ε, θα πρέπει να έχουμε ενίσχυση του ρυθμιστικού φορέα, να έχουμε επαρκές ε, δυναμικό. Ε, Παρ' όλα αυτά είμαι κατά ενός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις πρακτικές από τις διάφορες χώρες. όσον αφορά τους... Ε, όσον αφορά την ε, απελευθέρωση των ε, η Κομισιόν θα υποβάλει ένα τέταρτο πακέτο το οποίο θα έχει σημαντικές συνέπειες και δεν θα περιορίζεται μόνο στο σιδηρομικό τομέα μπορώ να επικροτήσω την ενίσχυση ε, των ε, ρυθμιστικών φορέων ε, και μπορώ επίσης να συμφωνήσω με τις διάφορες τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές συνθήκες. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός δεν επιτρέπει να οδηγεί σε κοινωνικό ντάμπινγκ και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου και την εποπτεία των συνθήκων εργασίας. Όλες οι προσπάθειες ε, που έχουν να κάνουν με την ε, χρηματοδότηση με βρίσκουν σύμφωνο. Και η απόρριψη των κατεξουσιοδότηση πράξεων επίσης με βρίσκει σύμφωνο. Μπορώ επίσης να συμφωνήσω με τις ε, τροπολογίες που ασχολούνται με την εσωτερική του εξωτερικού κόστους. Ίδιες συνθήκες για όλους τους τρόπους μεταφορών, για να αποφύγουμε στρέβλωση του ανταγωνισμού τους επόμενους μήνες θα πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε ώστε να εξετάσουμε επαρκώς τις ε, συμβαστικές τροπολογίες που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νταμτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Γκρός προηγουμένως αποκατέστησε αυτό που είναι η φιλοδοξία μας πριν από 10 χρόνια για το σιδηρόδρομο. Ξεκίνησε το εργοτάξιο, αλλά το εργοτάξιο παντού όπως συντίθεται. Τι απολογισμό μπορούν να κάνουν σήμερα οι εκλογές μας, οι Ευρωπαίοι πολίτες, πως εν γέννη το άνοιγμα δεν μεταφράστηκε ακόμα σε βελτίωση των υπηρεσιών. Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου σήμερα μάλιστα υπάρχει οπισθοδρόμηση των υπηρεσιών. Κοιτάξτε τι γίνεται σήμερα ανάμεσα στι διάφορε επιχειρήσει του σιδηροδρόμου ε, κοιτάξτε τι ανταγωνισμό κάνουν. Ε, ε, κάποιες φορές για λίγα ευρώ και θα δούμε ότι εκεί που τρένα ήταν διεθνή εδώ και πάνω από έναν αιώνα σήμερα ε, μεταφέρουν τον κόσμο μέσα σε ένα πούλμαν για να πάνε από το εθνικό τρένο Α στο τρένο Β γιατί δεν υπάρχει πια σύνδεση ανάμεσα στα δύο συστήματα. Απέναντι στους συμπολίτε μας δηλαδή τι κάνουμε, τους, ε, Κοροϊδεύουμε. Εγώ χαιρετίζω την εργασία και το θάρρο τη εισηγήτρια. Όποια και αν θα είναι η λύση την οποία θα καταλήξουμε, τώρα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για να Έχουμε αίσια έκβαση, αν θέλουμε, όπω το είπαμε και στην προηγούμενη συζήτηση και όπω το θύμισε και ο Ντομινίκ Κρικέ, να έχουμε μεταφορές επιταβών που να καταναλώνουν όσο γίνεται λιγότερο άνθρακα και νομίζω πως η Σιδηρόδρομη ακριβώς είναι τέτοια λύση. Είμαστε θύματα διαρκώ αυτό το θεσμικό όργανο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαρκώ κυνηγάμε τα συγκρούσει συμφερόντων. Εδώ λοιπόν οι συγκρούσει συμφερόντων σε διάφορα επίπεδα μπλοκάρουν το συμφέρον των συμπολιτών μας. Thank you very much. Before I bring in the Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν, να πω και εγώ ότι πιστεύω ότι ο Αντιπρόεδρος ε, Ρικέ ε, πολύ σωστά αναφέρθηκε στο που θα γίνουν οι πραγματικές μάχες για το θέμα αυτό. Ε, σίγουρα θα καταλήξουμε σε έναν ε, συμβιβασμό, θα έχουμε μια θέση του Κοινοβουλίου, αλλά η πραγματική μάχη θα γίνει με το Συμβούλιο, διότι όπως υπόθηκε, το Συμβούλιο ήδη έχει προσπαθήσει να αραιώσει, να αποδυναμώσει την πρόταση της Κομισιόν. Άλλωστε αυτό συνηθίζουν να κάνουν. Και όμως θα αντιμετωπίσουμε μία ε, σημαντική μάχη ε, στην προσπάθειά μας ε, προώθηση των σιδηροδρόμων. Αρχίζω και αμφιβάλλω αν, αν τα κράτη-μέλη θέλουν να προωθήσουν τις σιδηροδρόμους. Δεν νομίζω, ότι, νομίζω ότι κάποια κράτη-μέλη δεν θέλουν ευρωπαϊκό σύστημα σιδηροδρόμων. Είναι πολύ ικανοποιημένα εντός των δικών τους ε, συνόρων. Και έχουμε δει ε, τα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια να οχυρώνονται πάλι πίσω από τα εθνικά του σύνορα. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους. Και ναι, θα έχουμε κάποιες διαφωνίες, ε, θα ε, πρέπει να συζητήσουμε αν θέλουμε αποσύνδεση ή όχι, αλλά ε, νομίζω ότι η οχι αλλα νομιζω οτι η εκκληση προς τα κράτη-μέλη είναι τελικά ότι το status quo, η κατάσταση ως έχει, το να μείνουμε εδώ που είμαστε δηλαδή δεν αποτελεί λύση, δεν αποτελεί επιλογή. η ε, πρόοδος που έχω δει στις οδικές μεταφορές τα τελευταία χρόνια ε, ξεπερνάει κατά πολύ ε, τις ε, ε πρόοδους που έχουμε δει στους σιδηροδρόμους. Ε, δεν ε, προχωράμε με την ταχύτητα ε, τρένου ΤΕΖΕΒΕ, των ε, υπερταχείας. Πού βρισκόμαστε λοιπόν τώρα, πού θέλουμε να καταλήξουμε όσον αφορά ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα. Εάν εμείς εδώ εντός του Κοινοβουλίου δεν μπορούμε να θέσουμε τις προτεραιότητες ε, και τις αρχές για ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα, τότε σίγουρα με απόλυτη βεβαιότητα δεν θα ε, καθορίσει κάτι τέτοιο ούτε το Συμβούλιο των Υπουργών, διότι δεν τους ενδιαφέρει. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να στηρίξουμε την εισηγήτρια. Φυσικά θα υπάρξουν διαφωνίες, χρειαζόμαστε όμως μία σαφή θέση του Κοινοβουλίου όταν ψηφίσουμε τον Οκτώβριο και προχωρήσουμε τελικά σε αυτό που εγώ θεωρώ την πραγματική μάχη. Η πραγματική αυτή μάχη θα διεξαχθεί όπως πάντα με τα κράτη-μέλη που έχουν οχυρωθεί εντός του Συμβουλίου των Υπουργών. Ο κύριος Καστελέτη, εκ μέρους της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Φυσικά είναι αναπόφευτο να, το, να ξεκινήσω χωρίς να αναφέρω τις εξελίξεις της ε, προηγούμενης εβδομάδας. Παρά την πολύ συντηρητική θέση κάποιων κρατών μελών, ε, το Συμβούλιο τελικά κατέληξε να υιοθετήσει με μεγάλη πλειοψηφία την ε, γενική του θέση. Το κείμενο αυτό σίγουρα δεν είναι το ιδανικό, είναι αποτέλεσμα μακρών συζητήσεων ε, συμπεριλαμβάνουν πολλούς συμβασμούς, δεν ικανοποιεί απόλυτα την ε, Κομισιόν, διότι πολλές ε, διατάξεις έχουν αποδυναμωθεί, έχουν αραιωθεί, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει αλλάξει το πνεύμα Τη πρόταση τη Κομισιόν. Ε, η Κομισιόν ε, θέλει να ενθαρρύνει το Κοινοβούλιο να προχωρήσει γρήγορα. Σήμερα παρατηρούμε ότι σήμερα το πρωί αποφασίσατε να αναβάλλετε τη συζήτηση και την ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή σας. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι πριν ένα χρόνο, ε, κύριε Πρόεδρε, εσείς ε, στείλατε επιστολή στην Κομισιόν εκφράζοντας την ε, έκπληξη και την απογοήτευσή σας σχετικά με τις καθυστερήσεις στην υιοθέτηση της πρότασης της Κομισιόν. Θεωρήσατε ότι βρισκόμαστε υπό την πίεση της Επιτρέψτε μου να τελειώσουμε. Όχι κύριε, βρίσκεστε στην δική μου επιτρεπή εντός του δικού μου κοινοβουλίου. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Ε, λέει ο, ο κύριος Κομισιόν. Δεν θα πρέπει η Κομισιόν να κάνει διάλεξη στην Κομισιόν σχετικά με την ταχύτητα ε, της πρότασης μας για τους σιδηροδρόμους στη στιγμή που περιμέναμε χρόνια την πρόταση της Κομισιόν. Αυτό είναι το θέμα κλειδί. Προτείνω λοιπόν ότι αν αυτό είναι το ύφο της απάντησής σας μπορούμε να τη συντομεύσουμε και να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η Κομισιόν, είμαστε απογοητευμένοι με την απόφασή σας ε, για την αναβολή και αυτό μπορεί να διακυβεύσει την ε, πρόταση της Κομισιόν εντός επόμενης χρονιάς. Έχουν υποβληθεί πολλές τροπολογίες από τα μέλη της ε, Επιτροπής Τράν. Είναι όμως πολύ δύσκολο να εκφράσουμε τη θέση μας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Επιτρέψτε μου να πω όμως ότι κάποιες από αυτές αποδυναμώνουν ακόμα περισσότερο την πρόταση τη Κομισιόν, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν ε, το άρθρο 13 πολύ περισσότερο από ότι αποδυναμώνουν την ε, πρόταση τα κράτη-μέλη που ε, ε, υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Όσον αφορά την αποσύνδεση, έχει συζητηθεί το θέμα αυτό, δεν θα παραλάβω αυτά που έχουν υποθεί. Και επίσης η Κομισιόν είναι ανοιχτή απέναντι σε κάποιες προτάσεις κάποιες τροπολογίες σε μελών της Επιτροπής σας, αλλά αυτές που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών ρυθμιστών μας βρίσκουν ε, διάφωνους. Οι προτάσεις αυτές έχουν να κάνουν με την ικανότητα λήψη αποφάσεων ε, και άλλα. Θα ήθελα να τονίσω ότι το θέμα του ρυθμιστικού φορέα είναι ένας από τους βασικούς ε, στόχους αυτής της αναδιατύπωσης. Και η δυνατότητα δημιουργίας ε, ρυθμιστικού φορέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί μια δυνατότητα. Ε, πιστεύουμε όμως ότι θα πρέπει να βασιστούμε στο δίκτυο υπαρχών των ρυθμιστικών φορέων. Επίσης, πολλοί ευρωβουλευτές προτείνουν κάποιες εξαιρέσεις, παρεκκλήσεις. Αυτό είναι ευαίσθητο το θέμα οι παρεκκλήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν βάσιμους λόγους και να είναι περιορισμένες. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι όπως γνωρίζετε η αναδιατύπωση αυτή ε, στοχεύει στην κωδικοποίηση ε, των προηγούμενων προτάσεων. Ε, η Κομισιόν ε, έχει προσπαθήσει να τροποποιήσει μόνο κάποια μέρη ως αποτέλεσμα της διοργανικής συμφωνίας του 2001. Αυτή ήταν η προσέγγιση που υιοθετήθηκε και από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Προτού να δώσω το λόγο στον εισηγητή, να θυμίσω στην Επιτροπή ότι βρισκόμαστε σε μία νομοθετική διαδικασία και ε, είναι απαραίτητο να υποβληθούν τροποποιήσεις, ε, αν είναι απαραίτητο να ε, υποβληθούν τροποποιήσεις στην αρχική νομική πρόταση, ε, αυτό θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ε, νομοθετική διαδικασία. Η Επιτροπή μας ε, έχει την αρμοδιότητα να υποβάλει οποιαδήποτε τροποποίηση στην πρόταση της Κομισιόν εάν θεωρεί αυτό απαραίτητο και ειλικρινά είμαστε εκλεγμένοι από το λαό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μας κάνετε μάθημα για τη δημοκρατία. Η κυρία Σαρικιάνη παρακαλώ. <coughs> Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ε, όσους πήραν το λόγο και που ξεκαθάρισαν και τις ε, θέσεις. Όμως από ένα επίσημο, ένα μάλλον τυπικό θέμα το οποίο ανέφερε ο κύριος Κράμε, θέλω να ξεκινήσω, γιατί πιστεύω πως εδώ πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και πρέπει να έχουμε με βέβαιο σεβασμό ε, στη δουλειά που κάνουμε. Εγώ δεν νομίζω πως δεν ήμουν συνεργάσιμη, αλλά μπορώ πάντοτε να βελτιωθώ. Πάντως, δεν υπάρχουν προτάσεις συμβιβαστικές διαφορετικές από αυτές που στάλθηκαν σήμερα σε όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Την περασμένη εβδομάδα συναντηθήκαμε με τους εισηγητές και συμφωνήσαμε ότι ήταν δικό μου έργο να υποβάλω συμβαστικέ προτάσει σε σχέση με του εθνικού ρυθμιστικού φορεί, τη χρηματοδότηση και τι κατεξοδότηση πράξη και έπρεπε να τι υποβάλω πριν από την επόμενή μα συνάντηση που ήταν αύριο το πρωί, που προγραμματισμένη για αύριο το πρωί. Φτάσαν λοιπόν τα συμβαστικά κείμενα. Δεν υπάρχουν άλλα. Γι' αυτό θα ήθελα να υπάρχει σαφήνεια στη σχέση μας. Τώρα, αν πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο και καλύτερα, φυσικά και είμαι στη διάθεση όλων. Ε, θα το συζητήσουμε και αύριο, σίγουρα. Στην πρόταση αυτή νομίζω πως έχω συμπυκνώσει ωστόσο τις παρεμβάσεις πολλών, για, κυρίως όσον αφορά το πρόσωπο του ρυθμιστικού του ρυθμιστή που να θα είναι βέβαια ενισχυμένο ε, σε συμφωνία με τους όσους που με προηγήθηκαν, τον κύριο Κούν, τον κύριο Κρός, τον κύριο Τρεμόζα, όλους όσους δηλαδή τόνισαν πως ήταν ε, μια αρχή με δυνατότητες ε, συγκεκριμένες και αρμοδιότητες συγκεκριμένες καθώς και με ανεξαρτησία. Επίσης είναι πολύ είναι δυνατόν να βρεθεί μια λύση και πάνω σε αυτό δουλεύω όσον αφορά τις ενδείξεις για τα άρθρα 31 και 32 η κυρία Ζιλ. Η θέση τώρα που ανέφεραν ορισμένοι και ο κύριος Κράμερ σε σχέση με την ανάγκη του να περιμένουμε την ε, απόφαση του ΔΕΚ. Το Κοινοβούλιο, ωστόσο, πιστεύω ότι πρέπει να ασχολείται με τα νομοθετικά, ε, τις νομοθετικές προτάσεις είτε με τον αδονομοθετή. Δεν μπορούμε να αφήνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να... Ε, προσαρμόζει τις απόψεις του στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό πρέπει να είναι έργο δικό μας και το λέω με λίγη πικρία και στον κύριο Βίλσε ε, γιατί εγώ κατάλαβα ότι οι ευρωβουλευτές είναι εδώ για να αντιπροσωπεύουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Από τη στιγμή που εμείς, ε, αν ήμασταν εδώ για να αντιπροσωπεύουμε βιομηχα... Ε, εθνικές εταιρείε, επιχειρήσεις, τότε μάλλον κάτι δεν έχω καταλάβει καλά. Άμα είναι εδώ ο κύριο Βέλης για να αντιπροσωπεύει την Deutsche Bahn, ε, την Deutsche Bahn, ε, λυπάμαι, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αντιπροσωπεύουμε εδώ τους Ευρωπαίους πολίτες όλους. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και τις προτάσεις μου. Εν περιπτώσει, με πικραίνει κάπως αυτή η θέση, αλλά είμαι βεβαία ότι πρόκειται για παρεξήγηση, για λάθος. Συμφωνώ για τη θέση, με τη θέση του κυρίου Γκρός και ο οποίος νομίζω συνόπισε πολύ καλά ποιος είναι ο στόχος μιας μορφής ε, διαχωρισμού που να μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, ανεξαρτησία και να μην υπάρχουν διακρίσεις ε, στην πρόσβαση στο σιδηροδρομικό σύστημα. Είναι ενδιαφέρουσα και η πρόταση του κυρίου Αλκαντράουη, κυρίως όσον αφορά την απελευθέρωση. Είναι πολλές οι προτάσεις που γίνονται ε, από τον κύριο Καντσάν και άλλους, νομίζω πως από αυτού θα πρέπει να γίνει συζήτηση στο εσωτερικό της Επιτροπής Μεταφορών, ξεκάθαρη και ανοιχτή. Και ίσως θα μπορούσα να καλέσω την κυρία Ντουρά να διαβάσει πιο προσεκτικά το σχέδιο που υπέβαλα, καθώς και τις τροπολογίες που υπέβαλα, γιατί νομίζω πως η γραμμή αυτή είναι ξεκάθαρη. Αν δεν είναι, Είμαι έτοιμη να το ξεκαθαρίσω. Πιστεύω ωστόσο ότι εκεί είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και η συμμετοχή σε προηγούμενες συζητήσεις που έγιναν εδώ σίγουρα θα είχε ξεκαθαρίσει καλύτερα τη δική μου θέση, αν την είχατε ακούσει καλύτερα. Τώρα, όσον αφορά τη διατήρηση των κοινωνικών ρυθμίσεων. Συμφωνώ με την κυρία Τικάου. Εγώ θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντική η κοινωνική πρόνοια και έλαβα υπόψη όλες τις παρατηρήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τώρα, όσον αφορά την ανάγκη να μπορούμε να έχουμε μια αναδιατύπωση που να είναι πρόταση από πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου θαραλέα, πιστεύω πως αυτό είναι καθήκον των Ευρωβουλευτών να κάνουν μια πρόταση θαραλέα που να ξεπερνά τις λιγοστές φιλοδοξίες της Κομισιόν κυρίως, καθώς Η δουλειά που μας περιμένει το 2012 είναι πολύ δεσμευτική και αφορά το σιδηροδρομικό σύστημα και εδώ ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια, αποφα... μια αποσαφήνιση από τη στιγμή που αυτό το σιδηροδρομικό σύστημα είναι το σύστημα όπου πιστεύουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον. Κοινοβούλιο και Κομισιόν, γιατί είναι πιο οικολογικό και γιατί είναι αυτό που απαραίτητο θα πρέπει να βελτιωθεί και να ανοίξει. Αλλά και γιατί χρειαζόμαστε υποδομές από τα κράτη μας. Αν όντως αυτό θέλουμε, εντάξει. Διαφορετικά θα μείνουμε αφού ένα σχέδιο, ένα διατύπωση, και θα ξεκινήσουμε ούτε καν τις επόμενες σημαντικές ε, μάχες στην απελευθέρωση και τα όσα μας περιμένουν για το 2012. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν σαφήνεια σε σχέση με την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε σχέση με τις προτάσεις που μας φτάνουν από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ επαναλαμβάνω ότι το γεγονός ότι καθυστερήσαμε την ψηφοφορία και την αναβάλαμε για τον Οκτώβριο, μας δίνει περισσότερο χρόνο να το σκεφτούμε ε, μέχρι τον Αύγουστο και ε, μέσα στον Αύγουστο μάλλον και ελπίζω πως αυτό θα οδηγήσει τον εισηγητή, αφού θα την εισηγητρία αφού συνομιλήσει με όλους τους κοιόδης να καταλήξει σε κάποιες ε, συμβιβαστικές τροπολογίες και έπειτα, όπως είπα, προσβλέπουμε στην ψηφοφορία την Επιτροπή τον Οκτώβριο για να περάσει από την Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Επόμενο σημείο στην ελληνική διάταξη είναι η συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό. δίνω το λόγο στην κυρία Τικάου. Σίλβια. Σίλβια, μου επιτρέπεις δύο λεπτά ε, να πω ότι οποιοδήποτε αποχωρεί παρακαλώ ησύχω. Ησύχω. Μία συνεδρία επιτρέπεται σε κάθε αίθουσα του Κοινοβουλίου και αυτής προηγούμε εγώ. Οποιαδήποτε άλλο, άλλη συνεδρίαση πρόκειται να γίνει να βγει εκτός αιθούσης. Και παρακαλώ για σεβασμό προς την εισηγήτρια σας να ξεκινήσει την παρουσίαση της. Παρακαλώ Σίλβια. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συζητούμε σήμερα μια έκθεση για την απόφαση του Συμβουλίου προς τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διακόπτει μιλήτρια. Σύναψη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ του Μεξικού σχετικά με ορισμένε πτυχέ των αεροπορικών υπηρεσιών. ή διεθνεί σχέσει μεταξύ κρατών μελών και τρίτων κρατών διέπονται παραδοσιακά από διμερεί συμφωνίε στο μέτρων αεροπορικών υπηρεσιών. Ωστόσο, το 2002 το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι οι παραδοσιακέ ρήτρε περί καθορισμού αερομεταφορέα που περιέχονται στι διμερεί συμφωνίε αεροπορικών μεταφορών των κρατών μελών παραβιάζουν το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άρα επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, διαπραγματευτεί τη συμφωνία αυτή, η οποία αντικαθιστά ορισμένε διατάξει φυστάμενε 13 διμερεί συμφωνίε αεροπορικών μεταφορών που συνήθισαν μεταξύ 100 μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των ΗΠΑ του Μεξικού. Η συμφωνία αυτή έχει σημαντικέ ε, πτυχέ, εκ των οποίων το άρθρο 2 έχει να κάνει με τον καθορισμό του αεροματοφορέου, το άρθρο 2 την ασφάλεια, το 4 τη συμβατότητα με κανόνε ανταγωνισμό. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η αρχική συμφωνία που ετέθησε ισχύ το Μάιο του 2008 περιλάμβανε μια αμοιβαία διάταξη μια διάταξη αμοιβαιότητα που επέτρεπε τη φορολόγηση των καυσίμων για τι πτήσει εντό Ευρωπαϊκή Ένωση και τι πτήσει μεταξύ του Μεξικού και άλλων Αμερικανικών χωρών. Δυστυχώ όμω το Συμβούλιο δεν την απεδέχθηκε, τελικά αποσύρθηκε αυτή από το τελικό κείμενο. Η συμφωνία υπογράφηκε στι 15 Δεκεμβρίου του 2010, δεν εφαρμόζεται προσωρινά για να παραταθεί η εν λόγω συμφωνία, το Συμβούλιο χρειάζεται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εγώ είμαι υπέρ τη σύναψη ε, τη ολοκλήρου συμφωνία αυτή. Θα ήθελα να σα δώσω κάποια επιπλέον στοιχεία για να εξηγήσω την, ε, τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεξικού. Η συμφωνία αυτή. Το Μεξικό καταρχά είναι μια μεγάλη αγορά για του αερομεταφορεί Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι έχουν περίπου 2,5 εκατομμύρια επιβάτες το 2009 και 90.000 στόλους εμπορεύματα. Μεταφέρει στο Μεξικό. Ιδιαίτερα δεν θα ήθελα να υπογραμμίσω την ε, θέση του Μεξικού ως εμπορικού εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 21ος εμπορικός εταίρος και μεγάλη αγορά εξαγωγών μετά τις ΗΠΑ της Αμερικής και μάλιστα και πριν από την Κίνα. Για δε το εμπόριο των εμπορικών αγαθών, η αξία των εισαγωμένων από το Μεξικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση αγαθών είναι της τάξης των 9,9 δισεκατομμυρίων και των εξαγωμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Μεξικό της τάξης των 15,9 δις ευρώ. Τα σημαντικότερα εισαγόμενα προϊόντα είναι εργαλειομηχανές, οφθαλμολογικός εξοπλισμός και εξαγωγές, εργαλειομηχανές, ηλεκτρικός εξοπλισμός, χημικές ουσίες και μεταλλεύματα. Δεδομένες λοιπόν τη σημασίας αυτών των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και Μεξικού και του όγκου που εκπροσωπώ αυτέ οι δύο αγορέ, συνιστώ στην Επιτροπή μα να εγκρίνει την σύναψη της εν συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσω, να δώσω το λόγο ε, στους Ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, και την εισηγήτρια ε, για την δουλειά που έχει κάνει ε, στο θέμα αυτό. Πράγματι το Μεξικό είναι σημαντικός εταίρος ε, για μας ε, και ε, πάντα μου κάνει εντύπωση το πώς ε, πετυχαίνουμε καλύτερα αποτελέσματα με ε, χώρες που δεν είναι τόσο ισχυρή όσο είναι οι Ηνωμένε Πολιτείες. Και σημαντική είναι η συνεργασία την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, ε, ακολουθούμε εδώ μία καλή κατεύθυνση, την οποία ενδεχομένω να μπορέσουμε να ε, προχωρήσουμε πιο πέρα στο μέλλον. Ε, πάντως σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη βάση. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ την κυρία Τιτσάου για την έκθεση. Είναι άλλη μια από τις εκθέσεις στον χώρο των αερομεταφορών που συνάπτουμε, κάποιες συγκεκριμένες πτυχές των αεροπορικών ε, υπηρεσιών που ε, θίγει αυτή η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, που άλλωστε αποδεικνύει και τη μεγάλη σημασία του Μεξικού και πιστεύω θα πρέπει να ε, να γνωρίσουμε τη μεγάλη σημασία αυτού του εμπορικού εταίρου και να προχωρήσουμε και σε ευρύτερες ενδεχομένω συμφωνίες. Συχνά μιλάμε για Ηνωμένε Πολιτείε ε, και Καναδά. και Καναδά. Εγώ προτιμώ τον Καναδά ω καλό παράδειγμα, γιατί έχει μια πολύ πιο ισορροπημένη πολιτική σχέση με, με την Ηνωμένη Ευρώπη και γι' αυτό πιστεύω ότι θα ήταν καλό να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Καναδά στην περίπτωση του Μεξικού. Και άλλωστε πάντοτε έχουμε ε, προς υπογράψει του είδους ε, συμφωνίες λόγω των θετικών στοιχείων τους και το, ε, του γενικότερου συμφέροντος που εξυπηρετούν. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με την ασφάλεια των μεταφορών και με την εξυπηρέτηση των ε, επιβατών, την καλή λειτουργία των αερομεταφορών. Άρα πρέπει να την υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Τιτσάου. Συμφωνώ με το είπε κυρία Τιτσάου. Και προφανώς λαμβανωμένο εις υπόψη τη σημασία των εμπορικών σχέσεων που έχουμε τη χώρα αυτή, εκ μέρου της ομάδας μου υποστηρίζω την σύναψη της συμφωνίας. Καλώς. Κομισιόν, ο κύριος Μπουλκαβονή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την κυρία Τιτσάου για την έκθεση, τα συμπεράσματα και την σύσταση να εγκρίνει το Κοινοβούλιο τη συνάψη τη συμφωνίας. Που όπως υπενθύμισε η κυρία σε στόχο έχει να αναζωογονεί στην ασφάλεια δικαίου για αυτές τις 12 ε, διμερείς συμφωνίες που είχαν χαρακτηριστεί ε, παράνομες δυνάμει του ευρωπαϊκού δικαίου κατόπιν τη περίφημη εκείνη αποφάσεω του 2002 για τι εμπορικέ σχέσει με τι ΗΠΑ που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έτσι λοιπόν κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση αερομεταφορέα θα μπορεί να αναπτύσσει διαδρομέ μεταξύ οποιοδήποτε κράτου μέλου και του Μεξικού, εφόσον βεβαίω υπάρχει η σχετική διμερή συμφωνία και εφόσον υπάρχει και η, εφόσον είναι απελευθερωμένη η σχετική διαδρομή ελεύθερη διαδρομή. Το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως ξέρετε, πλέον τηρείται σε όλους τις στάσεις. Πρόκειται για την 45η σχετική συμφωνία, που έχει και την ιδιαίτερη σημασία της, γιατί όπως υπογραμμίσατε και εσείς κυρία Τιτσά, και όπως είπαν και οι κυρίες και κύριοι βουλευτές που έλεγαν το λόγο, αποτελεί μια δυνάμει βάση για να προχωρήσουμε προς κάτι το πιο σημαντικό, που θα μπορούσε να είναι φερειπίν μια γενική συμφωνία όπως αυτή που που διαπραγματευθήκαμε με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Βραζιλία με τη σύμπραξη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν λάβουμε υπόψη την εμπορική σημασία και τη σημασία της διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών, γιατί 2.600.000 επιβάτες ε, το χρόνο στο Μεξικό δεν είναι μικρή υπόθεση και αν κοιτάξουμε και το χάρτη, το παγκόσμιο χάρτη και τη θέση της Αμερική της Αμερικανικής Υπήρου, προφανώς η σύναψη μιας συμφωνίας με χώρα όπως το Μεξικό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σημασία γενικότερα. Προφανώ αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρόκειται να το μελετήσουμε περαιτέρω. Υπάρχουν δύο, όπω γνωρίζετε, προποθέσει. Καταρχά, η χώρα εταίρο να έχει και ίδια συμφέρον, ενδιαφέρεται και ίδια για τη σύνοψη μια ευρύτερη ε, συμφωνία, πράγμα το οποίο δεν γνωρίζουμε για την περίπτωση του Μεξικού. Και δεύτερη προπόθεση, ω συνήθω, το Συμβούλιο να δώσει τη σχετική εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορώ από εδώ να απευθύνω την ευχή να εκπληρωθούν και οι δύο αυτοί όροι. Και αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, με και έχω το λόγο, να, θα ήθελα να υπογραμμίσω απλώ προ την Επιτροπή σα ότι την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου των Μεταφορών, το Συμβούλιο ε, έδωσε εντολή διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εμπορικέ σχέσει με την, με την Μολδαβία, χώρα τη άμεση γειτονία, με την οποία μπορούμε να προχωρήσουμε τουλάχιστον σε διαπραγματεύσει ενώπιση συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία είτε εγώ είτε ένας από τους αντιπροέδρους όσον αφορά την ε, Μολδαβία. Η ψηφοφορία για το Μεξικό θα πραγματοποιηθεί τέλη Αυγούστου και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ την εισηγήτρια. Στα διάφορα εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Υπάρχει κανείς άλλος που έχει κάτι. Εάν όχι, να σας θυμίσω ότι... Ε, η επόμενη συνεδρία θα γίνει στις Βρυξέλλες 11 ε, Ιουλίου στις 3 η ώρα. Να σας ευχαριστήσω, ιδιαίτερα όσους άντεξαν όλο το απόγευμα. Και ο Πρόεδρος ε, ευχαριστεί ευγενικά και τους και εμείς ευχαριστούμε.